Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ, έχουμε αργήσει λίγο και έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα να συζητήσουμε σήμερα το πρωί. Πολλοί ευρωβουλευτές ε, εδώ την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχαν σε μια ακρόαση στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου όπου συζητήσαμε την ε, κρίση του ιού έμπολα και τον τρόπο αντιμετώπισης του. Στη συζήτηση αυτή λοιπόν ήταν ξεκάθαρο ότι επιγόντως πολύ γρήγορα πρέπει να αναλάβουμε κάποια δράση για να αντιμετωπιστεί ο ιός που σκοτώνει τόσους ανθρώπους και καταλήγει να είναι η πιο σημαντική κρίση σήμερα και πρέπει επίσης να πάρουμε και μαθήματα από την κρίση αυτή. Να δούμε λοιπόν τι κάνουμε σήμερα και τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια και μακροπρόθεσμα επίσης τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξανασυμβεί το ίδιο. Τα νούμερα είναι φοβερά ανησυχητικά γιατί πέθαναν πολύ περισσότεροι από αυτή την τελευταία κρίση παρά συνολικά από ότι Προηγουμένω από, πριν από 15 χρόνια που πρωτοεμφανίστηκε ο ιός μέχρι την τελευταία αυτή κρίση. Θα ακούσουμε για την έβολα λοιπόν σε λίγο για τον ιό αυτό. Προηγουμένως να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ένα θέμα έχουμε, εντάξει, συμφωνείτε όλοι. Τις ανακοινώσεις θα τις κάνω μετά. Για την ακρόση της επόμενης εβδομάδας θα τα ακούσετε και από τους συντονιστές σας έτσι κι αλλιώς. Οπότε ας περάσουμε ευθύ αμέσω στο θέμα μας αυτό για τον ιό έμπολα. Έχουμε εδώ διάφορους εμπειρογνώμονες από τις χώρες που έχουν πληγεί πρώτα απ' όλα τόσο άσχημα από τον ιό αυτό. Έχουμε εκπροσώπους από χώρες εταίρους που βοηθούν στην αντιμετώπιση του ιού. Έχουμε μη κυβερνητικέ οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται επί τόπου. Λοιπόν, θα ακούσουμε πρώτα απ' όλα τους εμπειρογνώμονες από τους ανθρώπους που πάνε στις χώρες αυτές. Στη συνέχεια μπορείτε να τους υποβάλλετε ερωτήσεις και στη συνέχεια θα ακούσουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που θα μπορέσουν να απαντήσουν στις διάφορες ερωτήσεις αλλά και στα σχόλια που θα έχουν ακουστεί προηγουμένως από τους εμπειρογνώμονες. Στο πάνελ έχουμε πρώτα απ' όλα την εξοχότητά του τον Ιβραήμ Σόρι, που είναι ο πρέσβης της Ιέρα Λεόνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Έχουμε επίση τον εκκληστικό διευθυντή, τον κύριο Λέον Κόκ, της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Είναι εδώ? Ναι. Ναι. Είναι, βλέπετε, μικρή αίθουσα, δεν έχουμε αρκετό χώρο για να έχουμε εδώ μπροστά όλους τους ομιλητές μας. γιατροί χωρίς σύνορα που βρίσκονται στις χώρες που έχουν πληγεί από τον ιό. Ο κύριος Στόκ από την, Επιτροπή, από την Οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ναι. Και μετά είναι ο κύριος Λεόν Πρόπτ, ο οποίος είναι του Ερυθρού Σταυρού. Είναι εδώ. Ο κύριος Ρίτσαρντ Μπράνον, διευθυντής της ανθρωπιστικής ε, βοήθειας από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στη Γενέβη και έχουμε και τον κύριο Κονζάλες από την USAID που είναι από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Την προηγούμενη εβδομάδα είπαν ότι θα στείλουμε μια μεγάλη ανθρωπιστική αποστολή στην πληγήσα περιοχή. Θα τα ακούσουμε και από εσά λοιπόν μετά. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτούς τους πέντε πυρογνώμονε πρώτα απ' όλα. Μετά μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας και στη συνέχεια θα ακούσουμε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΟ, ΕΦΚΟ και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράση Αρχίζουμε με του ειδικού μα στο θέμα. Μην ξεχνάτε, παρόλο που έχετε Ε, λίγο χρόνο, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξέρουμε εσείς τι χρειαζόσαστε, εμείς οι ευρωβουλευτές, τώρα αμέσως τι πρέπει να γίνει, αλλά και μακροπρόθεσμα τι μέτρα πρέπει να λάβουμε προκειμένου να μην ξαναέχουμε τέτοια κρίση η έμπολα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν η εξοχότης του, ο Ιβραήμ Σόρι, ο πρέσβης της Ιερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 8 λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είμαι εδώ, σε εκεί ο έδαφος, γιατί και εγώ ήμουνα βουλευτής στη χώρα μου για πολλά χρόνια. Πολλοί ε, βουλευτές εδώ γνωρίζουν και τους δικούς μας βουλευτές στα πλαίσια συνεργασίας. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εξοχότητες, ε, κύριοι πρέσβεις, αξιότιμοι, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής αυτής, αξιότιμοι συμμετέχοντες κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να εκφράσω την μεγάλη μου εκτίμηση και τις ευχαριστίες μου προς την Επιτροπή σας που οργάνωσε τη σημαντική αυτή συνάντηση για να ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά την επιδημία του ιού έμπολα στην λεκάνη του ποταμού Μάνου. Ιδιαίτερα μάλιστα στη χώρα μου, τη Σιέρα Λεώνα, αλλά και τη Λιβερία και την ε, Γουινέα. Η συνάντηση αυτή βέβαια δείχνει πόσο μεγάλη σημασία δίνει η διεθνής κοινότητα και ιδιαίτερα η ευρωπαϊκή κοινότητα και η εταίροι στην ανάπτυξη σε σχέση με το ξέσπασμα του ιού έμπολα και τις επιδημίες αυτής. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ επίσης για την εκλογή σας στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Κάποιοι από εσά ε, εκλεγήκατε για πρώτη φορά, άλλοι ήσασταν εδώ και προηγουμένως. Από τότε λοιπόν που αναγνωρίστηκε η επιδημία στη Σιέρα Λεώνα, τον Μάιο που μας πέρασε, μετά από την επιδημία στην Γουινέα τον Μάρτιο και στη συνέχεια και στη Λιβερία, η κυβέρνηση μαζί με τους εταίρους μας στην ανάπτυξη άρχισε να κινητοποιείται προκειμένου να διαθέσει πόρους για να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. Στα πλαίσια Αυτά λοιπόν η κυβέρνηση δημιούργησε ένα συντονιστικό μηχανισμό μαζί με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, μαζί με τους γιατρούς χωρίς σύνορα, την UNICEF και άλλα διεθνή σώματα. Επίσης δημιούργησε και μια διυπουργική επιτροπή για να κινητοποιηθούν τα Υπουργεία, διάφορα τμήματα και υπηρεσίες της χώρας και να οργανώσουν μια πρωτοβουλία έξι μηνών, μια στρατηγική για να αντιμετωπιστεί η επιδημία και να ληφθούν ό,τι έκτακτα μέτρα πρέπει να ληφθούν για να περιοριστεί και να ελεγχθεί η εξάπλωση της επιδημίας. Έπειτα, το ξέσπασμα και η αντίδραση σε αυτό από 60 μέχρι 90 μέρες ήταν κάτι που έγινε σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, τους γιατρούς χωρίς σύνορα και άλλες διεθνείς οργανώσεις, με αποτέλεσμα καλύτερη συνειδητοποίηση και αντιμετώπιση των ε, οικονομικών αναγκών για να πετύχει το σχέδιό μας. Επίσης κηρύχθηκε έκτακτη ανάγκη στη δημόσια υγεία τον Αύγουστο, κάτι το οποίο μας οδήγησε στο να απομονώσουμε κέντρα όπου ήταν παρόν ο ιός, να περιορίσουμε τις δημόσιες συγκεντρώσεις, να εισαγάγουμε νέα μέτρα όσον αφορά τις ταφές και επιπλέον να λάβουμε μέτρα για να συνειδητοποιήσει περισσότερο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και αυτό μέσω των τοπικών αρχών, θρησκευτικών ηγετών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, κοινωνίες των πολιτών, μουσικών, γυναικών στις λαϊκές, εμπόρων και μέσα ενημέρωσης. Ένα σημαντικό στοιχείο για τον έλεγχο της ασθένειας είναι βέβαια η εποπτεία και η αποφυγή των ε, κοντινών επαφών. Ιδιαίτερα δεδομένου ότι στην χώρα μου οι επαφές αυτές, οι προσωπικές, οι στενές επαφές είναι πολύ συχνές και συγκεντρώσεις πολύ κόσμου κοντά. Καταρχήν, τρεις από τις τέσσερις χώρες, εκτός δηλαδή από την ακτή ελεφαντοστού που βρίσκονται στην λεκάνη του ποταμού Μάνο, έχουν ε, πληγεί. Θελήσαμε λοιπόν να αναλάβουμε από κοινού δράση στα πλαίσια του MRU και της ECOVAS, οργανώνοντας μια διάσκεψη κορυφής την 1η Αυγούστου του 2014 και μεταξύ άλλων συμφωνήσαμε για μέτρα όχι μόνο για τη διαχείριση και τον περιορισμό της ασθένειας, αλλά και για να αποφύγουμε την εξάπλωση του ιού σε διεθνές πια επίπεδο και αυτό το κάναμε με ελέγχου κατά την έξοδο από τα σύνορα και τα αεροδρόμια. Αυτά βέβαια απαιτούν τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας για να καταπολεμηθεί η επιδημία και η εξάπλωσή της. Και υπήρξε βέβαια κάποια θετική αντιμετώπιση με οικονομικά μέσα, ιατρικά και οργανωτικά. Παρόλα αυτά, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε υποστήριξη γιατί η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι τεράστια. Μετά λοιπόν τη διάσκεψη, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ιερα Λεώνα ανέλαβε βήματα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στην ε, διάσκεψη και από του. Αναπτυξιακού μα εταίρου ω εξή. Πρώτον, να ενισχύσουμε τη δυνατότητα που έχουν τα διάφορα ιατρικά κέντρα προσφέροντας περισσότερες κλίνε, προσωπικό και εξοπλισμό. Δεύτερον, ενισχύοντας την ικανότητα των εργαστηρίων να κάνουν δοκιμές και να ελέγχουν δείγματα. Τρίτον, δώσαμε επιπλέον ασθενοφόρα και άλλα οχήματα και οργανωτική στήριξη. Τέταρτον, δώσαμε περισσότερο προσωπικό εξοπλισμό προστασίας και φάρμακα. Πέπτον, προσλάβαμε, αλλά οργανώσαμε και κατάρτιση για επιπλέον ε, προσωπικό στο τομέα της υγείας και έκτον ενισχύσαμε την δυνατότητα τηλεφωνικών κέντρων SOS. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, κυρία Πρόεδρε, η κυβέρνηση της Ιερα έλαβε έκτακτα μέτρα και ζήτησε από τον κόσμο να παραμείνει στα σπίτια του για τρεις μέρες ώστε να γίνει καλύτερα η ανείχνευση, ο έλεγχος και η εποπτεία. Στόχος του περιορισμού αυτού που εμείς το λέμε όζε του όζε είχε ως εξή. Θέλαμε να πετύχουμε 100% ενημέρωση και πληροφόρηση στα νοικοκυριά. Η κοινότητα να αποδεχθεί τους ασθενούντες από τον έβολο, ιδιαίτερα τα παιδιά. Να προωθήσουμε επίσης την πλήση των ε, χεριών και μοιράσαμε 1,5 εκατομμύρια σαπούνια. Επίσης θελήσαμε να ακτιθεί εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας και να ενισχύσουμε και τον έλεγχο μεταξύ κοιτώνων. Παρόλο λοιπόν το γεγονός ότι όλες οι δραστηριότητες της κυβέρνησης έχουν να κάνουν με τον έβολο, παρόλα αυτά υπάρχει κλιμάκωση στον αριθμό των ατόμων που νοσούν και των ατόμων που χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας ε, της ασθένειας αυτής. Δεν γνωρίζουμε καλά πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και σίγουρα η κατάσταση αυτή πλήττει και την οικονομία αλλά και όλο τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος φοβάται, δεν μπορεί να καταλάβει πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια ασθένεια η οποία σκοτώνει ανθρώπους, που εμποδίζει τους ανθρώπους να θάψουν τους δικούς τους, να μην μπορεί να αντιμεταπιστεί. Η κρίση έχει επιδεινωθεί και ο ιός αυτός δυστυχώς βρίσκεται πάντα ένα βήμα πριν από τις δικές μας τις δυνατότητες να τον αντιμετωπίσουμε. Έχουμε 1745 συγκεκριμένες περιπτώσεις που ξέρουμε, που έχουν χάσει τη ζωή τους δηλαδή. Μάλλον, ε, ατόμων που έχουν εμολυνθεί από τον ιό και 505 περιπτώσεις θανάτων που έχουν επιβεβαιωθεί. Η φύση τέτοια του ιού απαιτεί η υψηλή κατάρταση στο όλο το ιατρικό προσωπικό. πολλές ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία δεν έχουν πάντα τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και πολλά από αυτά τα δρήματα έχουν κλείσει. Οι διεθνείς κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση το ξέρουν ότι εμείς έχουμε αναμειχθεί σε δραστηριότητες ειρήνευσης και έχουμε πετύχει πολλά πράγματα όσον αφορά τους θεσμούς μας, τη βελτίωσή τους, την δημοκρατική διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου, την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα δικαιώματα της γυναίκας στη χώρα μας. Η απόσυρση της δύναμης του ΟΗΕ, της UNIPSIL τον Μάρτιο που μας πέρασε, μετά από την ε, επιτυχία της χώρας μας, είναι μια απόδειξη της βελτίωσης αυτής. Όμως δυστυχώς η οικονομική κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη προκειμένου να με τον ιό. Παρόλο που ο πληθωρισμός έχει μειωθεί, έχει φτάσει 6,5% τον Απρίλιο από 12% που ήταν τον ε, Δεκέμβριο του 2012. Η ανάπτυξη επίσης βελτιώνει φτάνουμε το 8%. Το Διαθέσιο Νομισματικό Ταμείο έχει επίσης πει ότι το ΕΠ θα πέσει 3,3% από 11,3% θα πάει στο 8%. Οι οικονομικές επιπτώσεις δηλαδή τους τελευταίους πέντε μήνες είναι τεράστιες. τα επιτεύγματα λοιπόν της χώρας στην περίοδο μετά τον πόλεμο δυστυχώς τώρα ανατρέπονται. Σε ολόκληρη τη χώρα οι επιπτώσεις της κρίσης αυτής γίνονται στιτές σε όλα τα επίπεδα ζωής. Και κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης, για τα σχολεία, τα γυμνάσια, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα γενικά παραμένουν κλειστά μέχρι δεν ξέρουμε πότε. Κύριε Πρόεδρε, η η Νέα και η είναι μέρος της διεθνούς κοινότητα και θέλουμε να συνεχίζουμε να παίξουμε το ρόλο που μας πρέπει στην παγκόσμια ατζέντα. Σήμερα αγωνιζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Ζητάμε λοιπόν από τις χώρες που έχουν επιβάλει ταξιδιωτικούς περιορισμούς και περιορισμούς της πτήση τους να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους και να βοηθήσουν έτσι τους ε, εργαζόμενους τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τους γιατρούς χωρίς σύνορα, να μπορέσουν να έχουν τη στήριξη που τους χρειάζεται. Δεδομένης της περιφερειακής φύσης ε, του ιού έμπολα, η πρέσβης Δυτικής Αφρικής εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά και της Αφρικανικής Ένωσης και των χωρών ΑΚΕ, έχουμε ξεκινήσει μια διπλωματία για τον ιό του έμπολα και κάνουμε έκκληση στους αναπτυξιακούς μας εταίρους να βοηθήσουν περισσότερο ιατρικά, οικονομικά, τεχνικά κλπ. κλπ προκειμένου να περιοριστεί και να εξαλειφθεί η επιδημία. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω την ευγνωμοσύνη της κυβέρνηση της Ιερά Λεόνε και της περιοχής για την αντίδρασή σα στο ξέσπασμα του ιού έμπολα που δώσατε 150 εκατομμύρια ευρώ και προηγουμένως 12 εκατομμύρια για να στηρίξετε τις ε, κυβερνήσεις των χωρών που επλήγησαν και να ενισχύσετε τις δομές υγείας με επιπλέον 38 εκατομμύρια από ένα νέο πακέτο. Και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί και μετά την αντιμετώπιση της κρίσης. Επιπλέον, επιπλέον επισητιστική βοήθεια Σα ζητάμε ε, νερό και σίγουρα η ανακοίνωση που έγινε στην συνάντηση της 19 Σεπτεμβρίου 2014 μας ενθαρρύνει με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που δήλωσε ότι επιπλέον 80 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν από τις χώρες μέλη για να συμπληρώσουν την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση του ιού έμπολα. Κύριε Πρόεδρε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε και όλους τους ευρωβουλευτές που συνεχίζουν να μας στηρίζουν κοινοβουλευτικά στην αντιμετώπιση του ιού έμπολα στην περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Σας κατευχαριστώ. Υπάρχει και ο πρεσβευτής Γκίνε εδώ τον οποίο ευχαριστούμε επίσης για την παρουσία του και είμαι βέβαιη ότι όλοι μας εδώ είμαστε αλληλέγγυοι με το λαό της χώρας, των χωρών σας που αντιμετωπίζει τόσο δύσκολες καταστάσεις. Και φυσικά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά. Σας ευχαριστούμε για αυτά που είπατε. Δεύτερος ομιλητής μας, ο κύριος Χριστόφορος Στόουξ από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και θα μας πει τι κάνει επιτόπου η οργάνωσή του και τι χρειάζεται ακόμα. Και εκείνος 8 λεπτά περίπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Είναι καλό το ότι έχουμε την... το κοινοβούλιο που σκύβει πάνω από αυτό το πρόβλημα. Θα σας ενημερώσω λοιπόν και θα σας πω το τι βλέπουμε επί τόπου, κάποια στοιχεία προβληματικά. Είναι σαφές λοιπόν πως ε, η κατάσταση είναι ακόμα εκτός ελέγχου και στις τρεις ε, χώρες που πλήττονται περισσότερο στη Λιβερία τώρα στην ε, Μονοροβία, η δυνατότητα ιατρικής βοήθειας δεν έχει αυξηθεί τους ε, τελευταίους μήνες και διώχνουν τον κόσμο από τα κέντρα υγείας σε μεγάλους αριθμούς, ξαναστέλνουν στα σπίτια τους ε, και δεν έχουμε και εικόνα για το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη χώρα, στις επαρχίες ε, εκτός ε, της Μονροβίας. Από όσο ξέρουμε υπάρχουν ελάχιστες κλίνες και δυνατότητες εκτός Μονροβίας. Στη Σιέρα Λεόν οι αριθμοί αυξάνονται όπως και στη Λιβερία και στην Αγουινέα μάλλον υπάρχει μια υποτίμηση του φαινομένου δεν υπάρχουν δυνατότητες παραδείγματος χάρη στη Freetown και τους στέλνουν στην άλλη άκρη της χώρας, στην ε, Κίνεμά ε, γιατί δεν ε, υπάρχουν κέντρα αντιμετώπισης της αρρώστιας τόπου. και για πρώτη φορά την τελευταία εβδομάδα φτάνουμε θα έλεγα ένα σημείο κορεσμού στην Κίνεμά και ανοίξαμε ένα καινούριο κέντρο στην Μπο στη Γουινέα όπου θεωρούμε πως ξεκίνησε η επιδημία πριν από 6-7 μήνες, εξακολουθούμε να βλέπουμε νέα ξεσπάσματα της επιδημίας σε διάφορα μέρη της χώρας, αν και η κατάσταση στην Κονακρή από ό,τι φαίνεται είναι υπό έλεγχο. Οπότε η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική για τις τρεις χώρες. Επίσης υπάρχει ανησυχία ε, για την πιθανή εξάπλωση σε γειτονικέ χώρες και τίθεται ζήτημα παρακολούθησης ε, στις μεθοριακές περιοχές, ειδικά σχέση με την ακτή του ελεφαντοστού. Όπως είπα λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο κορεσμού, διώχνουμε τους ασθενείς από τα κέντρα υγείας πίσω στο χωριό τους ε, και εκεί πέρα μολύνουν των πλησίων τους. Μέχρι στιγμής έχουμε εκθετική αύξηση, κάθε τρεις εβδομάδες διπλασιάζονται τα κρούσματα. Και έτσι έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα, το πότε θα γίνουν ε, οι λεγόμενες ε, αναπτύξεις ε, διαφόρων μέσων. Επίσης υπάρχει άλλη μια κρίση εντός της κρίσης. Κλείνουν τα νοσοκομεία σε πολλές από αυτές τις χώρες. Στη Μονοδοβία δεν υπάρχει ούτε ένα δημόσιο νοσοκομείο ανοιχτό σήμερα. Οπότε αν έχει κανείς μια κατάσταση η οποία μπορεί να μην είναι μοιραία, παραδείγματο χάρη ένα ανοιχτό κάταγμα, μπορεί να πεθάνει γιατί δεν ε, υπάρχει κάπου να πάει αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει και αυτή η κρίση μέσα στην γενικότερη κρίση. Λοιπόν, έχουμε πει πως είναι άνευ προηγουμένου η κρίση αυτή του τελευταίου εξαμήνου και υπάρχει θα έλεγα αρκετά μεγάλη ευαισθητοποίηση του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, Κίνας, Ιαπωνίας κτλ και μετά από έξι μήνες επιτέλους ε, έχουν γίνει κάποιες σοβαρές δεσμεύσεις που ανταποκρίνονται στο μέγεθος της κρίσης. Αλλά εάν έχουμε το χειρότερο σενάριο δεν αρκούν ε, τα πράγματα. Οι μίλησαν για 17 κέντρα με 17.000 κλίνες, λιγότερα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Γαλλία μάλλον κάπου στο, με ένα κέντρο αντιμετώπισης του ιού. Επιτόπου όμως δεν έχουμε δει τίποτα από αυτά ακόμα να λειτουργεί και ανησυχούμε πως ε, χάνουμε τη μάχη με το χρόνο κυνηγάμε την επιδημία όπως συνέβαινε εξ αρχής. Επίσης είναι σαφές πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να κινητοποιήσει τα κράτη-μέλη. Εμείς κάνουμε καθημερινές ενημερώσεις στα κράτη-μέλη. Ε, στη Γαλλία την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα αίτημα αυτή τη εβδομάδα από τη Γερμανία να τους ενημερώσουμε για να συζητήσουμε πώς μπορούν να στείλουν κάποια βοήθεια, τι εκπαίδευση χρειάζεται. Ε, αυτά γίνονται κατά περίπτωση όχι βάσει ενός συντονισμένου σχεδίου. Χρειάζεται όμως μια τριπλή αντιμετώπιση. Εθνική πόρη στις τρεις χώρες αυτές, αυτό γίνεται, αλλά όπως είπε και ο κύριος πρέσβης, πολλοί από τους ε, γιατρούς ε, και νοσηλευτές ε, ήταν τα πρώτα θύματα. Στα δικά μας τα κέντρα η μισή ε, ασθενείς ήταν ε, λιβεριανοί γιατροί και νοσηλευτές. Δύσκολο λοιπόν να αντιδράσουν. Οι ΜΚΟ αναπτύσσονται αλλά πάλι αρκετά αργά γιατί πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας και μετά όσον αφορά τον, ε, τη διεθνή κοινότητα έχουν γίνει ανακοινώσει, αλλά επί τόπου ακόμα δεν έχουν συμβεί πολλά πράγματα. Κάτι το οποίο θα θέλαμε να τονίσουμε είναι πως όλες οι δράσεις που αναλαμβάνονται πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την σοβαρή ε, ανάπτυξη, την, ε, με συγχωρείτε ασφαλή ανάπτυξη των ανθρώπων εκεί πέρα, με, να είναι σωστά εκπαιδευμένοι. Αλλιώ ε, θα βοηθήσουν ε, στην εξάπλωση της επιδημίας, γιατί είδαμε σε κάποιες αρχικές προσπάθειες το προσωπικό που πήγε να βοηθήσει να αμολύνεται. Ένα παράδειγμα, η ιατρική εκένωση που θα ήταν ε, κάτι εύκολο η απομάκρυνση των ασθενών ε, θα ήταν κάτι εύκολο να οργανωθεί. Ε, είχαμε απευθύνει επιστολή στην κυρία Άστον από τον Αύγουστο και Η δική μας είναι όλοι θέλοντες Έχουμε στείλει 350 άτομα μέχρι στιγμής ε, και ζητάμε τουλάχιστον να προταθεί μια λύση απομάκρυσης των ασθενών. Χρειάστηκαν πάνω από 48 ώρες για να προσγειωθεί ένα αεροπλάνο το οποίο έπρεπε να πετάξει από τις ΙΠΑ, Ήταν ευκολότερο, γρηγορότερο από ότι να έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν υπήρχε κάτι έτοιμο και ακριβώς αυτή η διαθεσιμότητα των μέσων ήταν κάτι το οποίο ζητούσαμε. Κάτι άλλο που νομίζουμε μπορεί να ε, γίνει εύκολα είναι μια αερογέφυρα για το προσωπικό και πιθανώς για τα δείγματα πιθανώς για μεταφορές ασθενών έγινε μια πρόταση προς την Κομισιόν να αναμένουμε απάντηση ε, η οργάνωσή μας και άλλοι φαντάζομαι κάνουν κάτι ανάλογο κάναμε την δικιά μας αερογέφυρα γιατί δεν μπορούσαμε να περιμένουμε άλλο μετά θέσατε το ζήτημα της ε, μακροπρόθεσμης ε, λύσης. Ε, χρειάζεται να υπάρξει προφανώς κάποια φαρμακευτική λύση και εμείς βεβαίως και άλλοι θα συμμετάσχουμε σε έρευνα επιχειρησιακή επιτόπου και βεβαίως εταιρείε και κυβερνήσεις πρέπει να προχωρήσουν πολύ πιο γρήγορα στην έρευνα πολύ γρηγορότερα από ό,τι συνήθως για φάρμακα και εμβόλια και πρέπει να αφιερωθούν περισσότεροι πόροι στην έρευνα και ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φαρμακευτική λύση και σαφώς πρέπει να γίνει μια προσπάθεια και να αφιερωθούν πόροι. Σήμερα η μόνη αντίδραση που έχουμε είναι το να στείλουμε ομάδες ε, επιτόπου πολλές και βεβαίως η αντίδραση επιτόπου των ε, κοινοτήτων εκεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Κάποια ανησυχητικά πράγματα ακούσαμε. Οπωσδήποτε βρίσκεται και η Κομισιόν εδώ και θα απαντήσει. Ξέρω πόσα ανησυχείτε. Τώρα, να δώσω τον λόγο στον κύριο Λεόν Προπ, αρμόδιο υπεύθυνο του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ερυθρού Σταυρού. Έχετε 6 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για τη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού. Θα σας κάνω μια γενική περιγραφή του πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και ποιες είναι οι προτεραιότητες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Από τον Μάρτιο φέτος δραστηριοποιηθήκαμε σε τέσσερις χώρες αλλά και σε εννέα άλλες όπου παίρνουμε προπαρασκευαστικά μέτρα για την πιθανή εξάπλωση της επιδημίας στο Τσάντ, στην Αφρικανική Δημοκρατία κλπ. και στη Γαμπία. Ως προς τα θεραπευτικά μέτρα στη Σιέρα Λεόν οργανώσαμε ένα κέντρο θεραπείας με 60 κλίνες στο κένεμα και ας μην μιλήσω για τα συγκεκριμένα θεραπευτικά μέτρα αλλά τα οργανωτικά. Διαχειριζόμαστε τους νεκρούς της Ιέρα Λεόνε, Λιβερία και Γουινέα γιατί όπως ξέρετε οι νεκροί ε, είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν γιατί είναι πολύ κολλητικοί. Σε μερικές χώρες όπως τη Γουινέα αναλαμβάνουμε πάνω από 95% των ταφών ώστε να είναι και αξιοπρεπής αλλά και ασφαλής και επίσης παίζουμε ένα ουσιαστικό ρόλο για την ε, παρεμπόδιση της εξάπλωση της ασθενείας. Υπάρχει βέβαια και το θέμα ψυχολογικής υποστήριξης μεταφοράς των ασθενών και όλες τις επιχειρήσεις των διεθνών οργανισμών που βρίσκονται εκεί τις έχουμε υποστηρίξει με 133 υπαλλήλους στο Σιέρα Λεόνε, Λιβερία, Γουινέα και Νιγηρία όπου εκπαιδεύσαμε 4.000 εθελοντές που μας βοηθούν και αυτοί. Τέλος, Είμαστε πολύ ενεργοί στην κοινωνική κινητοποίηση που θεωρούμε πολύ σημαντικό θέμα. 38 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από την ασθένεια και θα εκπαιδεύσουμε και άλλους εθελοντές για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Πριν από δύο εβδομάδες οργανώσαμε ένα φόρουμ για την πρόληψη στο Ντακάρ. Σε ε, υπήρξε κάλυψη από πολλά τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης και συμμετέσχων εκπρόσωποι και από τοπικά μέσα ενημέρωσης με στόχο να γίνει μια επίγουσα κοινωνική κινητοποίηση για να μπορέσουν να υποβοηθηθούν οι τοπικές αρχές να αντιμετωπίσουν την εξάπλωση και να περιοριστούν και τα αποτελέσματά της και κοινωνικά και οικονομικά πέρα από τα υγειονομικά μέσω καλύτερου συντονισμού και πληροφόρησης. Επίσης, να ακούσουμε τι μας λένε οι τοπικές κοινότητες οι ίδιες. Πρέπει να τις ακούσουμε. Οι συστάσεις από την διάσκεψη αυτή κατέληξαν στην κατάστρωση ορισμένων περιφερειακών προγραμμάτων και σχεδίων η roadmap η Αφρικανική Ένωση μας κάλεσε να οργανώσουμε μια ανάλογη διάσκεψη στην Ανατολική Αφρική για την ε, αντιμετώπιση της εξάπλωσης. Και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι ο αγώνας αυτός δεν θα κερδιθεί αν δεν καταφέρουμε να διαλύσουμε τους φόβους και την παραπληροφόρηση που κυκλοφορεί για το έμπολα, ώστε να μπορεί ο κόσμος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα πιο αποτελεσματικά γιατί η άγνοια δεν βοηθάει. Τώρα οι πόροι που χρειαζόμαστε προς στιγμήν δεν είναι αρκετοί. Μέχρι 30 εκατομμύρια έχουμε ζητήσει αλλά μόνο ένα τρίτο έχει καλυφθεί. Θέλουμε να αυξηθεί ο αριθμός των εθελοντών γιατί οι αριθμοί που διαθέτουμε δεν αρκούν καθόλου. Καταλαβαίνουμε ότι οι δωρητές θέλουν να αντιμετωπίσουν τα πράγματα κυρίως από υγειονομική άποψη θεραπευτική, αλλά αυτό δεν αρκεί για να σταματήσει η επιδημία. Πρέπει οι επίδοξοι δωρητές να λάβουν υπόψη τους όλες τις δραστηριότητες που να καλυφθούν και την κοινωνική κινητοποίηση και τις επαφές και την ψυχολογική υποστήριξη καθώς και capacity building η κατάσταση βέβαια είναι πολύ ρευστή και συνεχώς προσαρμόζουμε τα προγράμματά μας στις τρέχουσες ανάγκες και ζητούμε από όλους να είναι πολύ ελαστικοί. Τώρα η ασφάλεια της πρόσφατης εβδομάδες είδαμε ότι σημειώθηκαν πολλά προβλήματα ασφαλείας και ζητούμε από τις κυβερνήσεις, ιδίως ως προς τη μεταφορά από όλες τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν την ασφάλεια των εργαζομένων του Ερυθρού Σταυρού και των εθελοντών. Μας ανησυχεί πολύ η ασφάλεια των εθελοντών και του προσωπικού μας γιατί δουλεύουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και πρέπει να διασφαλίσουμε και την σωστή τους εκπαίδευση αλλά και την ασφάλειά τους καθώς και δυνατότητες ε, εκένωσης σε περίπτωση ιατρικού κινδύνου. Τέλος, ρωτήσατε ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες προτεραιότητες μας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να λυθούν τα βασικά προβλήματα μέσω μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων, δηλαδή και επένδυση σε υγειονομικές υποδομές και υπηρεσίες υγείας, αλλά χρειάζεται και η διανάπτυξη της δραστηριότητας τοπικών οργανώσεων και όπως του τοπικού Ερυθρού Σταυρού. Επειδή όμως περνάει ο χρόνος και χειροτερεύουν τα πράγματα, είναι πήγον να υπάρξει αντιμετώπιση τώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Επόμενος, Ρίτσαρτ Μπρέναν. Διευθυντής για την διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων στον ΠΟΗ στη Γενέβη. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ευκαιρία που μου δίνετε να πάρω το λόγο εδώ. Θα αναφερθώ και σε κάποιες παρατηρήσεις που έκαναν οι προλολήσαντες. Όπως υπόθηκε και νωρίτερα, η έκρηξη αυτή του ιού είναι κάτι άνευ προηγουμένου και λόγω μεγέθους και λόγω της γεωγραφικής εξάπλωσης. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο όπου να μπλέκονται πέντε διαφορετικές χώρες. Όσον αφορά τον εκθετικό τρόπο με τον οποίο αυξάνονται τα θύματα, είναι πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ σε έναν αστικό χώρο. Από τις 22 Σεπτεμβρίου έχουμε δει 5.800 περιπτώσεις με πολλούς θανάτους σε πέντε χώρες. Είναι περισσότεροι θάνατοι αυτοί από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα από όλε τις φορές που εμφανίστηκε ο ιός έμπολα κατά το παρελθόν μαζί. Έχουμε επίσης και περιπτώσεις θυμάτων μεταξύ του υγειονομικού προσωπικού. Οι μισοί μάλιστα έχασαν τη ζωή τους. Η πρόκληση λοιπόν που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστια. Έχουμε ένα σχέδιο, έχουμε μια στρατηγική, αλλά όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, δεν έχουμε τις ικανότητες ακόμα που χρειαζόμαστε πλήρως για να αντιδράσουμε. Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε. Τα Ηνωμένα Έθνη καθόρισαν στόχο που είναι βέβαια να σταματήσει η μετάδοση του ιού μέσα στους επόμενους ε, ξένα στόχοι οι οποίοι βέβαια έχουν να κάνουν με την μη μετάδοση πια του ιού. Πρόσβαση επίσης στις ιατρικές υπηρεσίες, όπως ακούσαμε πριν, πολλά νοσοκομικά ιδρύματα έχουν κλείσει. Όπως επίσης άλλος στόχος είναι νερό και τρόφιμα. Ένας άλλος στόχος είναι η σταθερότητα. Ακούσαμε τους κινδύνους. Εμείς θέλουμε οι κυβερνήσεις να παραμείνουν και να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στις χώρες αυτές. Οι στόχοι μας λοιπόν, αυτοί οι πέντε, είναι σαφείς και προσπαθούμε να τους πετύχουμε με τις δράσεις που έχουμε καθορίσει μέχρι τώρα. Χρειαζόμαστε όμως παραπάνω πόρους και σε χρήματα και σε ανθρώπινο δυναμικό. Οπότε λοιπόν και οι εταίροι μας έχουν κάνει διάφορα βήματα. Πρώτα απ' όλα φροντίζουμε να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε μέτρα ελέγχου της διάδοσης του ιού. Επιδημιολογικός δηλαδή έλεγχος, προκειμένου να παρακολουθούμε τις περιπτώσεις εμφάνιση του ιού καλύτερα. Έπειτα υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση στη θεραπεία. Είναι σημαντικά μέτρα αυτά προκειμένου να τηρούνται οι προδιαγραφές για την ταφή των θυμάτων, αλλά βέβαια και μέτρα ενημέρωσης του κοινού για να μην υπάρχουν προκαταλήψεις ή λάθος ενημέρωση. Δεν φτάνουν όμως αυτά. Πρέπει οι ιατρικές υπηρεσίες που έχουν σταματήσει να λειτουργούν να επαναλειτουργήσουν πρέπει, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, να έχουμε περισσότερες κλίνες για τους ασθενούντες. Γι' αυτό προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και άλλα συμπληρωματικά μέτρα. Να δούμε πώς η κοινότητα μπορεί να βοηθήσει και πώς η θεραπεία μπορεί να γίνει σε κοινοτικό επίπεδο και όχι μόνο στα νοσοκομεία. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε το θέμα και της υποθετικής διάδοσης του ιού σε άλλες χώρες και σε άλλες περιοχές. Γι' αυτό προσπαθούμε ε, να ζητήσουμε βοήθεια ώστε και οι γείτονες χώρες που δεν έχουν μέχρι τώρα παρουσία του ιού να προετοιμαστούν έτσι ώστε να αποφύγουν την είσοδο του ιού στις χώρες αυτές. Περιμένουμε τους επόμενους μήνες και άλλες χιλιάδες περιπτώσεις και μέχρι τον Νοέμβριο ίσως να έχουμε 20.000 περιπτώσεις ολόκληρη την περιοχή. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερες δυνατότητες επιτόπου και περισσότερο προσωπικό για να επανδρώσουν τα κέντρα θεραπείας του ιού πρώτα απ' όλα. Οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν το προσωπικό, στη Λιβυρία για παράδειγμα η Αμερικανική κυβέρνηση δεν στέλνει υγειονομικό προσωπικό στα κέντρα αυτά. Χρειάζεται όμως. Έχουμε ελάχιστους επίσης εταίρους που μπορούν να βοηθήσουν και στην περίπτωση των ε, θανάτων να στηρίξουν τις οικογένειες και να αποφύγουν τη διάδοση του ιού. Χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο για να ενισχυθεί επίσης το κυβερνητικό δυναμικό. Επιπλέον, έχουμε περιορισμούς προκειμένου να πείσουμε τους διεθνείς εταίρους να μας βοηθήσουν. Ακούσατε και από τους προλαλήσατες ότι είναι ανάγκη να μπορούν τα θύματα μάλλον τα θύματα που είναι μεταξύ του υγειονομικού προσωπικού, ανεξάρτητα από το ποια χώρα προέρχονται, από ποιο οργανισμό είναι, να μπορούν να μεταφέρονται από τις χώρες αυτές που πλήττονται από τον ιό έβολο και να μπορέσουν στη δικιά τους τη χώρα να θεραπευτούν. Να υπάρχουν άρα τακτικές πτήσεις από τις χώρες μας προς τις χώρες αυτές της Αφρικής ενώ πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν σταματήσει να πηγαίνουν. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι οι δομές των χωρών μελών. 3.000 στρατιώτες έχει διαθέσει η Αμερικανική κυβέρνηση. 500 μονάδες θεραπείας του Ιέμπολα έχει προσφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο στην ε, Σιέρα Λεόνε. Και υπάρχει και ανακοίνωση από τον ΟΗΕ για μια αποστολή ανταπόκριση στην διάδοση του ιού έμπολα, προκειμένου στις τρει χώρε που πλήττονται περισσότερο να υπάρχει παρουσία της μονάδας αυτής. Εφόσον υπάρχει καλός συντονισμός, θα περάσουμε από αυτό που κάνουμε τώρα που είναι να σταματήσει η διάδοση του ιού στις χώρες αυτές, να το δούμε γενικότερα και να σταματήσει η διάδοση του ιού πέρα από τις χώρες αυτές επίσης. Πέντε σημεία ακόμα. Πρώτα απ' όλα, αν δεν υπάρχει μαζική αντιμετώπιση, οι προκλήσεις που θα έχουμε για την μη διάδοση του ιού παρεπέρα δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί εύκολα. Ζητάμε λοιπόν από τις χώρες μέλη να συνεργαστούν μαζί μας, να προσδιορίσουν συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες θα πάνε στις χώρες που πλήττονται και σε συντονισμό με την Αμερικανική κυβέρνηση και εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου να μπορέσουν να βοηθήσουν επί τόπου. Χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο λοιπόν. Χρειάζεται επίσης οι χώρες μέλη να βοηθήσουν να μπορούν να μεταφέρονται οι από το υγειονομικό προσωπικό πίσω στις χώρες τους. Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει. Και εμείς ανησυχούμε λοιπόν που δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις μέχρι τώρα από αυτού και σας ζητάω να υπάρξει ένας τέτοιος μηχανισμός για την γρήγορη επιστροφή των ασθενούντων. Θέλουμε την αερογέφυρα επίσης, όπως ακούσαμε και πριν, και ενθαρρύνουμε τις χώρες μέλη και τους εταίρους μας τα Ενωμένα Έθνη, άπαξ και υπάρξει η αποστολή αυτή του ΟΗΕ και υπάρξει περισσότερο υλικό επιτόπου, να μην ξεχάσουμε ότι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εκεί είναι να σταματήσουμε τον ιό σε 6 με μήνες και να μην παρασυρθούμε και ασχοληθούμε περισσότερο με στρατιωτική οργάνωση και όχι με την καταπολέμηση του γιου αυτού καθεαυτού. Ευχαριστώ πάντως που μου δώσατε την ευκαιρία να πάρω το λόγο εδώ. Πρόεδρος, ναι, σημειώνουμε αυτά που λέτε την επίγον. Ξέρω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σημειώνει όλα αυτά και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Τελευταίος ομιλητής, ειδικό Ακούσαμε από τις χώρες, τον πρέσβη, ακούσαμε από τις οργανώσεις που είναι επιτόπου, ακούσαμε από εσά για το συντονισμό των προσπαθειών. Τώρα θα ακούσουμε έναν μετέρο που έχουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούσαμε 3.000 στρατιώτες σαν παριατρικό προσωπικό θα πάει. Ο κύριος Γκοζάλης λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για 6 λεπτά έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Good morning, Chairman McAvin and distinguished members. Καλημέρα σα, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα. Οι ΕΠΑ συμφωνούν με την αξιολόγηση του Κοινοβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα στο ψήφισμα του Στρασβούργου πως ε, η εμπολά αποτελεί μεγάλη <clears throat> αντιμετώπιση στην περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια. Σήμερα θα σας εξηγήσουμε την στρατηγική των ΕΠΑ και να τονίσω τέσσερις στόχους. Πρώτον, έλεγχος της επιδημίας. Δεύτερον, τα μακροπρόθεσμα, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Τρίτον, ενίσχυση της ε, υγειονομικής υποδομής και τέταρτον, μια ευρύτερη παγκόσμια αντίδραση και θα τονίσω πώς συνεισφέρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΠΑ ενισχύουν τις ε, προσπάθειές τους για να αντιμετωπίσουν το ξέσπασμα αυτό. Τον Αύγουστο η USAID έστειλε ειδικού από το Κέντρο Αντιμετώπισης ε, Ασθενειών, το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Υγείας ε, στην ε, Freetown και στη Μονοροβία. Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές, βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες και βεβαίω παρέχουμε βοήθεια η οποία σώζει ζωέ. Μέχρι στιγμή έχουμε εξοδεύσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια στην περιοχή και έχουμε δεσμεύσει άλλα 75 εκατομμύρια δολάρια. Έχουμε στείλει πάνω από 16 τόνους ιατρικού εξοπλισμού και στηρίζουμε και το πρόγραμμα τροφίμων του ΟΗΕ που ε, δίνει ψητιστική βοήθεια. Μαζί με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ, ΜΚΟ και λοιπούς προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε ιατρικό προσωπικό και προσωπικό επιμελητίας καθώς και ομάδες ασφαλούς ταφής. Ε, σκοπεύουμε μέχρι το τέλος του να έχουμε 300 κλίνες για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Ε, ο πρόεδρος Ομπάμα την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε μεγάλη αύξηση στη βοήθειά μας. Κατόπιν ετήματος της ε, Λιβερίας θα στήσουμε ένα στρατιωτικό επιτελείο με 3.000 προσωπικό μια προσπάθεια αρκετά μεγάλη συγκρινόμενη με αυτή της ITs με στόχο να ε, μπορούμε γρήγορα να διοχετεύσουμε προσωπικό και υλικό στην Δυτική Αφρική. Επίσης ε, θα συσταθεί ένα κέντρο εκπαίδευση όπου θα εκπαιδεύονται 500 άτομα τη βδομάδα και θα πάει και ένα νοσοκομείο εκστρατείας ε, του Υπουργείου Άμυνας στην Μονροβία το Υπουργείο Άμυνας θα διαθέσει για τον στόχο αυτό πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια. Όμως ε, δεν θα πετύχει η προσπάθειά μας, δεν θα είναι ολοκληρωμένη χωρίς μια ευρύτερη στρατηγική. Μέσω μιας εκστρατείας ενημέρωσης θα δώσουμε πληροφορίες στο πώς μπορούν να προστατευτούν οι άνθρωποι καθώς και 400.000 ε, σετ προστασίας. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Γουινέα σκοτώθηκαν 11 άτομα σε μια εκδήλωση ενημέρωσης. Ε, φαίνεται λοιπόν πως υπάρχουν ακόμα προβλήματα στην ενημέρωση. Για το λόγο αυτό επίσης στηρίζουμε τις ε, προσπάθειες εκπαίδευσης του κοινού μέσω μήνυμάτων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών στις τοπικές ε, γλώσσες, φυλαδίων, υπεθρίων διαφημίσεων και ενός τραγουδιού με ντόπιους μουσικούς τέλος τα Εθνικά Ιδρύματα Υγείας μας ε, αναζητούν αυτή τη στιγμή ένα εμβόλιο και ο πρόεδρος Ομπάμα ζήτησε από το Κογκρέσο 50 εκατομμύρια ε, δολάρια για να δοκιμάσουμε διάφορα υποψήφια φάρμακα και εμβόλια. Να σας πω τώρα το τι σκοπεύουμε να κάνουμε για τις επιπτώσεις στην περιοχή. Συζητάμε με τους ε, διεθνεί εταίρου μα για το πώς μπορεί να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην περιοχή. Έχουμε τέσσερις βασικούς στόχους. Διατροφική ασφάλεια, ανθρωπιστική προστασία, ενίσχυση της κυβερνητικής σταθερότητας όσον αφορά την παροχή βασικών υπηρεσιών και μείωση του οικονομικού αντικτύπου ενισχύοντας τη φορολογική ικανότητα των κρατών. Οι δωρητέ έχουν ήδη αναπτυξιακά προγράμματα εκεί πέρα και θα χρειαστεί κάπως να στραφούν προς αυτό το πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν κάποια βραχυπρόθεσμα ζητήματα, που μπορούν, κάποια βραχυπρόθεσμα πράγματα μπορούν να γίνουν αμέσω. Παρέχουμε ήδη ψητιστική βοήθεια, ε, τροφή και νερό, ειδικά στις απομονωμένες κοινότητες. Ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει διαθέσει 100 εκατομμύρια δολάρια προς Λιβερία και Σχέρα Λεόνε, κάτι το οποίο βεβαίω ε, θα ενισχύσει τη σταθερότητα. Ήδη υπάρχει μια παγκόσμια εκστρατεία για να αντιμετωπίσουμε τις συστημικές αδυναμίες του δημοσίου συστήματος υγείας στις περιοχές αυτές. Την Παρασκευή αυτή, οι Υπουργοί από 40 χώρες, 6 διεθνείς οργανισμούς και 5 περιφερειακούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο για να δεσμευτούν σε βάθος 5 ετίας ε, και σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις περιοχής για να αντιμετωπιστούν οι βιολογικές αυτές απειλές. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει μια δέσμευση εκ μέρους της παγκόσμιας κοινότητας έτσι ώστε εντός τριών ετών να μπορούν να ανοιχνεύουν και να αντιμετωπίζουν τέτοιες μολυσματικές απειλές όπως η έμπολα. Ελπίζουμε να συνταχθεί μαζί μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, να αναφερθώ στην ανάγκη συντονισμού των δωρητών. Οι ΙΠΑ πιστεύουν πως εδώ πέρα χρειάζεται ο ηγετικό ρόλος του ΟΗΕ και χαιρετίζουμε ιδιαίτερα το ότι ο Γενικός Γραμματέας όριζε τον Ντέιβιντ Ναβάρο για το θέμα αυτό και άρα θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 28 ε, Αυγούστου πρότεινε ένα σχέδιο δράσης για να κινηθούμε γρήγορα με τρόπο συγκεκριμένο. Αλλά οι μεγάλοι δωρητές όπως είπα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσουν τον ΟΗΕ με αυτή την φοβερή πρόκληση. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε εμείς ε, με την ε, Σόβας ε, Καναδά, Γερμανία, ΗΠΑ και Γαλλία οι βασικοί δωρητές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετική στον τομέα αυτόν. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναλάβει τον ηγετικό ρόλο στη Χέρα Λεόνε και η Γαλλία στη Γουινέα. Ενώ η ΕΠΑ έχει επικεντρωθεί στην Λιβερία. Έχουν επικεντρωθεί στην Λιβερία. Και βεβαίως με αυτό τον καταμερισμό εργασία και χρήση των πόρων. Όμως υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Πύρα και Γενεοδορία. Οπωσδήποτε χρειάζονται λεφτά, αλλά ο ΙΕ και οι γιατροί χωρίς σύνορα έχουν ζητήσει την αύξηση των δωρεών, ειδικά σε είδο, κάτι το οποίο δεν μπορούν να κάνουν οι ΜΚΟ. Θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία να δούμε πώ θα μοιραστούμε πόρου για αερογέφυρε και εκένωση ασθενών. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να διαβεβαιώσουμε όσου είναι επιτόπου και φροντίζουν πώ θα υπάρχει φροντίδα επιτόπου ή ε, ελήψη αυτού αερομεταφορά. Επίσης πρέπει να δούμε την εμπειρία που υπάρχει εντός της Αφρικής. Ε, χρηματοδοτούμε μία αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης για να σταλούν πάνω από 100 άτομα, γεωνομικό προσωπικό. Ε, διεθνής ε, στήριξη άρα με αφρικανική πύρα. Επίσης πρέπει να ενθαρρύνουμε την αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβερία να συνεχίσει την ειρηνευτική της αποστολή αν και οι χώρες αυτή τη στιγμή σκέφτονται να αποσύρουν τα στρατήματά τους λόγω της έμπολα. Πρέπει λοιπόν επίσης να υπάρξει και μία έγκαιρη προετοιμασία και περιορισμός της εξάπλωσης και να υπάρξει σαφής ορθή πληροφόρηση και να μην υπάρχει το στίγμα επίσης της ε, μόλυνσης. Επίσης να δούμε πώς θα κινητοποιήσουμε την διασπορά των χωρών αυτών. Τέλος, και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να στηρίξει περισσότερο τα όσα γίνονται και η ΜΚΟ οπωσδήποτε. Όπως είπε και ο πρόεδρος Ομπάμα, η κατάσταση θα χειροτερεύσει πριν καλυτερεύσει. Όμως έχουμε την ευκαιρία να σώσουμε πάρα πολλές ζωές και έχουμε ευθύνη να δράσουμε. Το οφείλουμε αυτό στους ε, θαραλέους γιατρούς και νοσοκόμους που παλεύουν εκεί πέρα κάθε μέρα και σε αυτούς που έχασαν ήδη τη ζωή τους. Οφείλουμε λοιπόν να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να σταματήσει αυτή η επιδημία και μαζί με την ε, Ευρώπη θα συνεργαστούμε για να καταπολεμήσουμε αυτή την απειλή στη διεθνή ειρήνη και τη σταθερότητα. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν όλους τους ομιλητές. Έδωσα και λίγο παραπάνω χρόνο γιατί θεώρησα ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε όσους έχουν επιτόπια εμπειρία. Και μόνο στο Σέφιλντ στην πόλη μου ξέρω ότι άκουσα ανθρώπους που έχουν πάει στη Σιέρα Λεόνε και ανέφεραν τις εμπειρίες τους και νομίζω ότι τέτοιου είδους πληροφόρηση είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, θέλω να αφήσω χρόνο και για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Κομισιόν. Μόνο τέσσερις συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ποιος άλλος ζητάει. για να δω πόσο χρόνο θα διαθέτουν. Έχω τους τέσσερις προηγούμενους. Κανείς άλλος. Ενρίκε Γκερέρο. Για να είμαστε βέβαιοι πόσο χρόνο θα έχουμε. Βέντα. Ο πρεσβευτής της Γουινέας, ναι. Μάλιστα κύριε. Πόσους έχουμε λοιπόν δέκα. Παρακαλώ λοιπόν ο καθένας δύο λεπτά. Και μετά αν υπάρξει χρόνος αφού ακούσουμε την Κομισιόν μπορούμε να επανέλθουμε. Δύο λεπτά ο καθένας λοιπόν. Τώρα μετά θα ακούσουμε τα όργανα και ύστερα μπορεί να επανέλθουμε. Στίαρ πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καθώς και όλους τους ομιλητές. Ιδιαίτερα εκφράζω την αλληλεγγύη μας προς τον πρεσβευτή, τους ευευτές της Γουινέας και της Ιέρα Λεόνε. Είχαμε μια χρήσιμη συζήτηση και ψήφισμα στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα. Δυστυχώς θα ξαναέρθει και την επόμενη φορά στην Ολομέλεια γιατί όπως ξέρουμε θα διπλασιαστεί μάλλον ο αριθμός των κρουσμάτων. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο μας είπε η Επίτροπος Γεωργίευα ότι δεν έχει υπάρξει κρούσμα από το διεθνές προσωπικό, αλλά τώρα ξέρουμε ότι υπάρχει ένα κρούσμα από τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Επίσης μάθαμε ότι χρειάζονται 48 ώρες για την εκένωση ενός ασθενούς με αεροπλάνο, γιατί πρέπει να έρθει αεροπλάνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά να πάει στην Ευρώπη. Αυτό χρειάστηκε για αυτήν την γιατρό λοιπόν. Άρα υπάρχουν ακόμη ελλείψεις μεταξύ και μεγάλο χάσμα μεταξύ υποσχέσεων και πραγματικότητας. Αν και υπάρχει πρόοδος δεν αρκεί. Από τις πληροφορίες μου ξέρω ότι τα υγειονομικά κέντρα από τους γιατρούς χωρίς σύνορα στα υγειονομικά αυτά κέντρα ξαναστέλνουν τους ασθενείς στα σπίτια τους γιατί δεν έχουν αρκετά μέσα. Να πηγαίνουν λοιπόν οι άρρωστοι, επιστρέφουν στα σπίτια τους, σημαίνει ότι διαδίδεται η ασθένεια. Και δεν νομίζω ότι έφτασε το ζενήθ της πολιτικής πίεσης που χρειάζεται για να υπάρξει η απαραίτητη αντίδραση. Στο ψήφισμά μας <coughs> της περασμένης εβδομάδας Ζητάμε συγκεκριμένα προγράμματα με προθεσμίες, αλλά πρέπει να δούμε και τι μπορεί να κάνει η δική μας Επιτροπή να ζητήσει περισσότερη πληροφόρηση κλπ. Θα μιλήσουν βέβαια και οι εκπρόσωποι της Κομισιόν και της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων, αλλά είναι ζωτικό να χρησιμοποιήσουμε όλο το πολιτικό βάρος που διαθέτουμε για να γίνει κάτι συγκεκριμένο από τις χώρες μέλη. Και τελικά, τέλος, θέλω να ξανατονίσω τη σημασία που έχει να ηγηθεί ο ΙΕ της προσπάθειας αυτής και να μην ε, υπάρχουν διαμάχες μεταξύ οργάνων και οργανισμών. Και εμείς να τον στηρίξουμε τον ΟΗΕ. Με αυτό τελειώνω. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ζάλτ Γκόριντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είμαστε ταχύτεροι από τον ιό και αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Ο ιός είναι ταχύτερος από μας και την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο είπαμε, τα είπαμε, αλλά αν χρειάζεται να προσθέσουμε ένα επιχείρημα για να χορηγηθεί τουλάχιστον 20% για τις βασικές υγειονομικές υπηρεσίες. Αυτό το αποδεικνύει η κρίση του ιού έμπολα. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους ε, προσώπους των οργανώσεων που με κίνδυνο της ζωής τους προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον έμπολα και τους γιατρούς χωρίς σύνορα και τον Ιρθρό Σταυρό και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τον ΙΠΑ που αποφάσισαν να στείλουν υλικό και στρατιωτικό. Για πρώτη φορά βλέπω τέτοια ανθρωπιστική ανταπόκριση με όλα τα μέσα και στρατιωτικά. Χρειάζονται 3.000 κλίνες προς στιγμήν. Γιατί σε δύο εβδομάδες ο αριθμός των κρουσμάτων θα έχει διπλασιαστεί. Αυτό δείχνει τι γεωμετρική πρόοδος υπάρχει. Καλό είναι βέβαια να γίνονται προβλέψεις για το μέλλον, αλλά πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο διαχειριστήκαμε την κρίση μέχρι τώρα και αυτό είναι σκάνδαλο. Εγώ είμαι υπέρ της πολυπλευρικότητας, αλλά έχω σκανδαλιστεί. Ποιος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, ποιος μας ανάγκασε να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων, κανείς. Δεν έγινε τίποτα σχετικά. Και τι έκαναν οι διεθνείς οργανώσεις, νομίζω ότι είναι μεν πρόημο να το πούμε, αλλά πρέπει να δούμε ποιος έκανε τι και πότε και ποιος δεν έκανε τίποτα. Ερωτώ λοιπόν και από την Κομισιόν. Μπορείτε να μας παριθμίσετε όλες τις ανταποκρίσεις, τις απαντήσεις, τις αντιδράσεις που ήταν είτε μηδενικές είτε καθυστερημένες λόγω έλλειψης σπόρων. Εγώ συνεννοούμε συχνά με επιστήμονες και ερευνητές και κάθε οργάνωση λέει ότι φταίει η άλλη. Δεν έχουμε λεφτά, είναι αργές οι διαδικασίες, μα οι διαδικασίες αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα της κατάστασης, γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα, δεν, δεν πρέπει να χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο και γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα υπάρχοντα μέσα. Ήδη έχουμε καταδικάσει στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για λιγότερο σοβαρά θέματα. Είναι μια ευκαιρία να κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη. Εγώ δεν δέχομαι πια να είμαστε βουβοί μάρτυρες μπροστά σε τέτοια σκάνδαλα. Όσο για τις εκενώσεις είναι ντροπή που η Ευρώπη δεν κατάφερε να οργανώσει μια τέτοια υπηρεσία που είναι μια Γαλλίδα γιατρός ή νοσοκόμος έπρεπε να περιμένει τέσσερις μέρες πριν να βρεθεί αμερικανικό τσάρτερ για να τη μεταφέρει στο Παρίσι. Είναι σκάνδαλο όλα αυτά. Το μόνο που με καθησυχάζει κάπως είναι ότι την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεχτήκαμε ένα από τα καλύτερα ψηφίσματα που δεχτήκαμε ποτέ και το συνυπέγραψα βέβαια και εγώ. Τουλάχιστον έτσι έγινε μια αρχή ρεαλιστικής αντιμετώπισης. Ευχαριστούμε. Στο τέλος, ίσως θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να ετοιμάσουμε μια επιστολή ή κάτι, να δούμε τι θα μας πει και η Επιτροπή. Μισελ Λιβαρή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ που οργανώσατε και αυτή τη συζήτηση στροκυλής τραπέζης κατά κάποιο τρόπο για τον Ιέμπολα. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Γκέρενς και εγώ και θέλω να πω μια που εδώ έχουμε όλους τους συνομιλητές παρόντες. 22 Μαρτίου μάθαμε. 23 Σεπτεμβρίου είναι σήμερα, 6 μήνες μετά. Μπορούμε λοιπόν πράγματι να αναρριτηθούμε. Πώς είναι δυνατόν να μας χρειάζονται έξι μήνες για να αποφασίσει σήμερα ο κύριος Ομπάμα να στείλει 3.000 στρατιώτες. Ο Επίτροπος μας είπε ότι η Επιτροπή έκανε τη δουλειά της. Ναι, αλλά η δουλειά της τελικά δεν ήταν στο ύψος των προσδοκιών που περιμένουν εδώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίζονται για την καταπολέμηση του ιού και για την οργάνωση των γιατρών χωρίς σύνορα. Είσαστε εδώ, θα σας τα πω. Έχω την εντύπωση ότι εσείς δεν ε, φωνάξατε το κατεπήγον την έκτακτη αυτή κατάσταση για να κινητοποιηθούν όλοι. Η οργάνωση αυτή που έχει τις δομές που μπορεί... Γιατί να μην ακουστεί νωρίτερα. Γιατί να είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε που λένε θα στείλουμε 3.000 στρατιώ, στρατιώτες. Ναι, στρατιώτες, έτσι, όχι ιατρικό προσωπικό. Αυτό όμως δημιουργεί πρόβλημα, γιατί αυτοί θα πρέπει να φάνε. Και γιατί όχι ιατρικό προσωπικό. Οι χώρες τι ζητάνε. Ιατρικό προσωπικό που θα καταρτήσει ιατρικό προσωπικό επιτόπου. Αυτό χρειάζεται. Δεν είναι ή εμείς που θα πάμε εκεί και θα πούμε στους αρρώστους πρέπει να κάνετε αυτό και εκείνο το άλλο εμείς οι λευκοί. Όχι, οι άνθρωποι επιτόπου θα μιλήσουν στους ασθενείς και θα τους πούνε τι πρέπει να κάνουν. Εμείς λοιπόν πρέπει να πάμε εκεί να βοηθήσουμε το ιατρικό προσωπικό επιτόπου για να βοηθήσει με τη σειρά του τον τόπιο πληθυσμό. Θέλω να ρωτήσω γιατί ε, Σιέρα Λεόνε, μια που έχουμε εδώ τον ε, πρέσβη. Στη Σιέρα Λεόνε λοιπόν απομονώσατε τον πληθυσμό για τρει μέρε, τον κρατήσατε στα σπίτια του. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, γιατί ήσασταν η μόνη χώρα που το είπε αυτό. Είπε τρει μέρε κανεί δεν θα βγει στον δρόμο. Αλλά οι ειδικέ ομάδε πηγαίνανε επί τόπου στα σπίτια, στα νοικοκυριά και ελέγχανε την κατάσταση. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Και μια που θυμάμαι την παρέμβαση των ΗΠΑ στην ΑΕΤ, λέω προσοχή, οι ντόπιε κυβερνήσει πρέπει να εμπλέκονται. Εγώ έχω συγγενεί στη Λιμπέρια, στη Λιβυρία και πηγαίνουν στα σπίτια. Όταν υπάρχει ένας ασθενής ή ένας νεκρός, δεν θέλουν να τον βγάλουν από το σπίτι. Οπότε εγώ ρωτάω εσάς, πείτε μου, τι πρέπει να κάνουμε. Όταν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όπως οι γιατροί χωρίς σύνορα που έχουν κάνει εξαίρετο έργο, πηγαίνουν στα σπίτια, τι κάνουν, πώς βγάζουν τους μολυσμένους από τα σπίτια χωρίς να μολύνουν και άλλους. και τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και πώς μπορεί να συνδυαστεί αυτό με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Λοιπόν, τώρα για το υγειονομικό προσωπικό μάθαμε για την ε, γυναίκα εκείνη που μολύνθηκε. Πώς όμως, γιατί δεν το λέτε. Αποτέλεσμα, δεν θέλει να πηγαίνει ο κόσμος εκεί επί τόπου. Πρέπει να ξέρουμε πώς δημιουργήθηκε η μόλυνση αυτή. Και η εκένωση αναφέρθηκε και εσύ σε αυτό. Και μένα με εκπλήσει πώς είναι δυνατόν να συνεδριάζουν οι Υπουργοί Υγεία, να τίθεται το θέμα της εκένωση και το να μαθαίνουμε ότι ένα Αμερικανικό στρατιωτικό αεροπλάνο πήγε και πήρε τη γυναίκα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερα για το συντονισμό μεταξύ χωρών μελών και για την αερογέφυρα. Πάντως για το κατεπήγον του συντονισμού, ναι, οι, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν έναν, μια οργάνωση για αυτή τη δουλειά να δραστηριοποιηθεί περισσότερο. Γιατί οι γιατροί χωρί σύνορα, εντάξει, μπορεί να μην μπορούν να κάνουν περισσότερα, αλλά με τι άλλο το καμπανάκι του συναγερμού έπρεπε να το έχουν χτυπήσει πολύ νωρίτερα. Έχουμε ένα P4. Ξέρετε, είναι ένα νοσοκομείο που μελετάει στην Καμπόν τον ιό και το έχουμε και στη Λιόν. Μα από το 1996 γνωρίζουμε το ιό έμπολα. Οι φαρμακευτικές εταιρείες τι λένε, δεν παράγουν φάρμακα γιατί δεν υπάρχει μεγάλο κέρδος. Μα δεν είναι δυνατόν. Θα έπρεπε να πούμε στα φαρμακευτικά εργαστήρια θα πάρετε χρήματα, δημόσιο χρήμα, αλλά θα φτιάξετε φάρμακα για την έμπολα. Γιατί τώρα είναι η αρχή, σήμερα είναι εκεί, μεθαύριο θα είναι αλλού. Ναι, όντως ξέρουμε αυτό πώς λειτουργεί και η Επιτροπή Περιβάλλοντος μπορεί να βοηθήσει. Λόλα Σάντζεθ τώρα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ όλους όσοι πήραν το λόγο εδώ γιατί μας εξήγησαν ποιες είναι οι ανάγκες αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Θέλω να ρωτήσω τον πρέσβη της Ιερα Λεόνε κάτι. Η αναπτυξιακή βοήθεια φυσικά παίζει σημαντικό ρόλο. Ενισχύει τις δημόσιες δομές των εταίρων μας. Τον ρωτάω λοιπόν, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην τήρηση των στόχων των αναπτυξιακών αυτών και τα επίπεδα στα οποία έχει φτάσει η επιδημία. Και άλλη ερώτηση προς τον κύριο Στόξ από την, τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Νομίζω ότι το έπαιξε κάθαρο ότι χρειάζονται τεχνικό εξοπλισμό, ε, χώρους για να γίνεται απομόνωση, ιατρικό προσωπικό, υγειονομικό. Πιστεύει ότι χρειάζονται πράγματι μικτές αποστολές στρατιωτών και πολιτών ή μόνο στρατιωτών. Γιατί είναι πολλά χρήματα. Καλό θα είναι να πηγαίνουν σωστά. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σύντομοι. Ο κύριος Πόγκα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι πήραν το λόγο εδώ σήμερα και που μας εξήγησαν το έργο τους ο καθένας. Και συγχαρητήρια και ευχαριστώ για τη δουλειά ακριβώ αυτή που κάνετε για να θεραπεύσετε τους ασθενούντες από τον έμβολο. Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω. Πρώτον, είναι αλήθεια ότι η διεθνής κοινότητα πήρε χρόνο για να αντιδράσει. Αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το είπαν και άλλοι φίλοι, πήρε μέτρα για να βοηθήσει τις χώρες που πλήττονται από την επιδημία. Δεύτερη παρατήρηση. Ο συντονισμός μεταξύ των διεθνών φορέων είναι κάτι αναγκαίο πια. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί οι δράσεις οι οποίες αναλαμβάνονται να είναι από συνοχή για να είναι και αποτελεσματικές. Τρίτη παρατήρηση. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη δράση μας για να αντιμετωπίσουμε την έκτακτη αυτή κατάσταση, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι χρειάζονται τα κατάλληλα μέσα στις πληγήσεις χώρες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τέτοια υγειονομική κρίση, δηλαδή ενίσχυση των υγειονομικών δομών, αλλά και χρηστή διαχείριση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Καθή Μπέρνταν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, προλαλήσαντες που μας περιέγραψαν ε, το τι συμβαίνει στη χώρα, στο μέτωπο, αν θέλετε, ε, με τους ανθρώπους που κινδυνεύουν καθημερινά. Και πρέπει να τους σκεφτόμαστε και να τους ευχαριστούμε. Έχω κάποιες ερωτήσεις το πληροφοριακό δελτίο που μας δώσατε φαίνεται πως πολλοί επιζούν. οι ασθενείς επιζούν. Ε, όντως γίνεται αυτό. Μετά, όταν επιζήσουν, έχουν ανοσία ή μπορεί να ξαναρωστήσουν. Και εάν ναι, τους χρησιμοποιούμε, γιατί αν έχουν ανοσία, μπορεί ε, να τους εκπαιδεύσουμε για να βοηθήσουν ε, τους άλλους. Το άλλο θέμα είναι η αστικοποίηση. Η δυσκολία με τον αστικό πληθυσμό είναι βεβαίως ο συγχρονισμός πολλών ανθρώπων σε λίγο χώρο. Και φαίνεται πως είναι αστική αυτή η αρρώστια. Κατόπιν, αυτό το οποίο είπε η Λίντα για τη διασπορά. Ξέρω πως ε, στη δικιά μου την περιφέρεια υπάρχουν πολλοί άνθρωποι από τη Δυτική Αφρική και θα ήθελα να μάθω πως μπορώ να τους κινητοποιήσω για να κάνουν κάτι. Επίσης απογοητεύομαι γιατί δεν βλέπω να υπάρχει σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. Ε, βασικά πράγματα δηλαδή αυτά. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Ξέρουμε πως ε, όλοι λέμε πως πρέπει να είναι η τελευταία αυτή επιδημία. Ε, λέμε πως ε, εντάξει χρειαζόμαστε το χύψη και ωμέγα τα οποία δεν υπάρχουν. Αερογέφυρα, απομάκρυνση ασθενών, ένας γιατρός ε, πήγε στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπήρχε από ό,τι φαίνεται μόνο μία μονάδα αρμόδια στο Λονδίνο. Και σε 15 μέρες, εντάξει, ανένυψε. Αλλά ε, είναι τρέλα αυτό. Ξέρουμε πως ε, αυτές οι ασθένειε υπάρχουν. Πραγματικά έχουμε μόνο μία, ξέρω, λίγες μονάδες απομόνωσης. Ε, θα έπρεπε να έχουμε και κάποιες μονάδες εκστρατείας για να τις στείλουμε εκεί ποιο είναι το σχέδιο της ε, Κομισιόν. Και εγώ οπωσδήποτε όλοι τους ε, συμπονάμε με αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ και Γκερέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω ένα γενικό σχόλιο, μια ερώτηση και μια πρόταση. Το γενικό σχόλιο είναι ότι όλοι οι ειδικοί που πήραν το λόγο εδώ, όλοι οι εκπρόσωποι από τα διάφορα όργανα και οργανώσεις, είπαν ότι δεν φτάνουν τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να αντιμετωπίσουν την επιδημία. Και εκθετικά οι ανάγκες αυξάνονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αλήθεια ότι αντέδρασε, αλλά αντέδρασε προσπαθώντας να δώσει οικονομικά μέσα τα οποία κανονικά ήταν για άλλη δουλειά. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να δεχτούν και να επικυρώσουν ένα έκτακτο ταμείο προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι έκτακτες ανάγκες. Η ερώτησή μου τώρα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δηλαδή στη διαχείριση της κρίσης. Γιατί γενικά μιλώντας όλες οι ανθρωπιστικές κρίσεις, το κύριο πρόβλημα που έχουν είναι την ενότητα των δράσεων, το συντονισμό ουσιαστικά των όσων βρουν επιτόπου. είναι στρατηγική σημασία χωρίς να στοιχίζει πολλά χρήματα. Και έρχομαι στην πρότασή μου τώρα. Η πρότασή μου έχει να κάνει με την κοινωνία των πολιτών. Σε ανθρωπιστικές κρίσεις, δυστυχώς, η καταστροφή γίνεται επιτόπου και δεν είναι πάντα εμφανής από τα μέσα ενημέρωσης. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, είχαμε δύο περιπτώσεις κρίσης έμπολα και όταν οι δύο αυτές περιπτώσεις έγιναν γνωστές, όλα τα μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν. Και μόλις έπαψε η κρίση, τελείωσε, εξαφανίστηκε το θέμα. Ένα λοιπόν από τα θέματα που θα πρέπει να κάνει η Επιτροπή μας αυτή είναι να κρατήσει ζωντανό το θέμα αυτό στα μέσα ενημέρωσης και παντού. Ίσως όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα μετά τη συζήτηση που είχαμε εκεί, οι συντονιστές με την Πρόεδρο να ζητήσουν από τα κράτη-μέλη σε σχέση με την αυριανή ε, διάσκεψη δωρητών στη Νέα Υόρκη. Η Επιτροπή Ανάπτυξης δηλαδή, έχοντας ακούσει τις διάφορες οργανώσεις που δρούν ε, επιτόπου, αξιολογεί την ανάγκη για περισσότερα μέσα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση και ζητάει από τις κυβερνήσεις των χωρών μελών μας αύριο στη Νέα Υόρκη να δεσμευτούν για επιπλέον χρήματα από αυτά που είχαν ε, μέχρι τώρα αποφασίσει να δώσουν. Αυτό γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Πρόεδρος, θα μας πούνε οι αξιωματούχοι που έχουμε εδώ ποια είναι τα σχέδια για την Νέα Υόρκη και για την επόμενη συνάντηση της Παρασκευής. Τελευταίος μιλητής από τους Ευρωβουλευτές, ο κύριος Βέντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ όλους τους εκπροσώπους των οργανώσεων που ήρθαν εδώ του ΟΗΕ, ΠΟΗ, γιατροί χωρί σύνορα κλπ. κλπ. Αυτά που ακούσαμε, τα στοιχεία που μας έδωσαν δεν είναι βέβαια πολύ ευχάριστα, μας δίνουν την εικόνα της κρίσης που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ο χρόνος πιέζει φυσικά και υπάρχουν σχέδια που έχουν αναπτυχθεί, προγράμματα κλπ. Αλλά φτάνουν πάντα με μεγάλη καθυστέρηση. Πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Στόξ. Γιατί από αυτά που άκουσα, κατάλαβα καλά, είπατε ότι δεν υπάρχουν φάρμακα για το έμπολα, έτσι. Τι σημαίνει αυτό για τις πληγήσεις χώρες και τι σημαίνει αυτό για μας. Είναι θέμα πολιτιστικό, νοτροπίας. Ξέρω ότι και κάποιοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν επί τόπου. Και προς την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Είχαμε και παλιότερα τέτοιες κρίσεις έμπολα το 2003 με υψηλή θνησιμότητα, 9%. Αλλά σταμάτησε η μετάδοση και η κρίση. Τώρα το ότι επανέρχεται ο ιός. Με τι έχει να κάνει. Έχει να κάνει με τις μεταφορές, έχει να κάνει με τον τρόπο αναμετάδοσης. Ο κύριος Μπρέναν είπε ότι σε λίγο δεν θα είναι περιφερειακή η κρίση, πολύ πιθανό να γίνει παγκόσμιο το πρόβλημα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Πριν να περάσουμε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, θα δώσω το λόγο στον ε, πρέσβη της Γουινέας. Συλλεγγύνα, τρία λεπτά, τέσσερα το πολύ, ε γιατί θέλουμε να ακούσουμε ξανά και τους προσκεκλημένους μας όλους. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν γιατί μας επιτρέπετε να συμμετάσχουμε σε αυτή την εκδήλωση. Λέγομαι ως Μανσίλα, είμαι ο πρέσβης της Γουινέας της Βρυξέλλες. Η Γουινέα προεδρεύει αυτή τη στιγμή των χωρών ΑΚΕ, 119 χωρών, και γι' αυτό εκφράζομαι και ως πρέσβης αλλά και ως προεδρεύων τον και για τους επόμενους έξι μήνες. Σε αυτά τα πλαίσια κυρία Πρόεδρε θα θέλαμε να συνδεθούμε και εμείς με εκδηλώσεις προσεχής του Κοινοβουλίου εδώ ή στο Στρασβούργο που να αφορούν αναπτυξιακά και υγειονομικά θέματα. Για τον έμπολα είμαι από χώρα που όπου και εκεί εξέσπασε η επιδημία το Μάρτιο και αμέσως η κυβέρνηση και ο αρχηγός της ε, πήραν δρακόντια μέτρα για να αντιμετωπίσουν την επιδημία. Ήρθαν οι γιατροί χωρίς σύνορα, εργάστηκαν εξαιρετικά. Όταν όμως βλέπουμε πώς εξαπλώνεται η επιδημία, από το Μάιο-Ιούνιο είχαν αρχίσει να λένε ότι ελέγχθηκε. Δυστυχώς από τον Ιούλιο-Αύγουστο όμως υπήρξε νέα έκρηξη. Στις γειτονικέ χώρες διευκολύνθηκε αυτό και από τα ταξίδια Σιέρα Λεόνε και Λιβερία και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή την ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση και για τις τρεις χώρες. Ο πρέσβης της Σιέρα Λεόνε που τον ευχαριστώ μίλησε εκ μέρους των ενδιαφερομένων χωρών και σας ανέφερε όλα τα μέτρα που λήφθηκαν και στη Λιβερία και στη Γουινέα και στη Σιέρα Λεόνε για να αντιμετωπιστεί ο ιός έμπολα. Και ευχαριστώ ειλικρινά τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους γιατρούς χωρίς σύνορα, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη Γαλλία που κινητοποιήθηκαν και τη Μεγάλη Βρετανία καθώς και όλες τις χώρες μέλη της Ένωσης που κινητοποιήθηκαν για να μας βοηθήσουν. Θεωρούμε ότι η διεθνής βοήθεια αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στην ταχύτητα που χρειάζεται και ο αρχηγός της κυβέρνησης της Γουινέας που είναι αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη μεθαύριο θα πάει σε μια διάσκεψη που οργανώνει ο Γενικός Γραμματέας Μπάν Κιμούν για το έμπολα. Σήμερα θα ακούσει για τις κλιματολογικές αλλαγές και μεθαύριο για το έμπολα. Εξ ονόματος λοιπόν των τεσσάρων χωρών θα δώσει περαιτέρω πληροφορίες για τα μέτρα που έλαβαν οι χώρες αυτές. Δεν υπάρχει βέβαια ούτε εμβόλιο ούτε φάρμακο και επομένως ο καλύτερος τρόπος αυτή τη στιγμή είναι η πληροφόρηση και η πρόληψη καθώς και η ενδυνάμωση των υγειονομικών υποδομών. Γι' αυτό η βοήθεια που χορηγούν οι διάφορες χώρες είναι κάτι για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες αλλά πρέπει και να ενισχυθεί. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Air France, το Royal Air Maroc, της Bruxelles Airlines που δεν σταμάτησαν τις μεταφορές και τα ταξίδια στις χώρες μας. Είναι γνωστό αλλά πρέπει να το ξαναπούμε να μην απομονωθούν οι χώρες αυτές. Το κλείσιμο των συνόρων και η απομόνωση δεν συμφέρει κανέναν, δεν βοηθάει κανέναν. Τέλος, για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, θα ήθελα εξ ονόματος των χωρών και 119 όπως είπα, να ζητήσω την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να οργανωθεί μια επίγουσα διεθνής διάσκεψη αλληλεγγύης στις Βρυξέλλες. Γίνονται προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας και το χαιρετίζουμε αυτό, αλλά πιστεύουμε ότι και ο έμπολα είναι ένα είδος τρομοκρατίας και ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση για αυτόν τον πόλεμο κατά της αρρώστιας αυτής. Κάνουμε λοιπόν μια έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να οργανωθεί σύντομα στις Βρυξέλλες όπως είχε γίνει άλλη φορά και για το Σαχέλ μια διεθνής διάσκεψη για τον έμπολα στην οποία να μπορέσουν να γίνουν γνωστοί τα στοιχεία από την κοινή γνώμη αλλά και να εκφραστεί περισσότερο η διεθνή αλληλεγγύη. Ακόμη μια φορά κυρία Πρόεδρε ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα όσα κάνει για να, υποστηρίξει, να στηρίξει τις χώρες μας και ελπίζουμε ότι με αυτή τη μελλοντική διάσκεψη η βοήθεια αυτή θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε βέβαια ανοιχτοί για οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να τεθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Οπωσδήποτε θα διαβιβάσουμε αυτά τα οποία μας είπατε στους συναδέλφους από την ΑΚΕ. Τώρα θα ακούσουμε τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος Σόρενσεν, Γενικός Διευθυντής ΕΚΟ. ΔΕΒΚΟ. δύο άτομα, δεν ξέρω ποιοι θα μιλήσουν. Κυρία Βερονίκ Λορέντσο και ο κύριος Ντιπιέ Βέρς και ο κύριος Πι... Πίτερης από την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν ξέρω αν θα μιλήσετε με μία φωνή. Χρήσιμο θα ήταν να το καταλάβουμε γιατί υπάρχει και θέμα συντονισμού. Ποιος είναι επικεφαλής, ο ΙΕ, ποιος συντονίζει. πρέπει να ακούσουμε λοιπόν το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τρία διαφορετικά πράγματα, εμείς κάνουμε αυτό και εμείς κάνουμε αυτό. Ε, μην μου τα πείτε τρεις φορές τα ίδια. Κύριε Σόρνσεν, τέσσερα λεπτά. Ε, ήταν πολλές οι ερωτήσεις, δεν ξέρω πόσο έχουν ε, και οι συναλφοί σας. Συντονιστείτε μεταξύ σας. Ε, κύριε Σόρνσεν, δεν θα αρχίσει τώρα ο συντονισμός κυρία Πρόεδρε, αλλά οπωσδήποτε από το Μάιο είμαστε σε συνεννόηση και ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχαμε καθημερινές ή μέρα παραμέρα επαφές βίντεο διασκέψεις με τις αντιπροσωπείες μας, ε, με την Σάρα, αλλά και με τους συναδέλφους της στην Ουάσιγκτον. Συντονισμός υπάρχει. Ξέρουμε το τι κάνουν ε, τα διάφορα, διάφορες υπηρεσίες και είναι συμπληρωματική η δράση μας. Ο καθένας έχει τη δουλειά του. Οπότε προχωράμε. Μία γενική παρατήρηση πρώτα απ' όλα. Είναι κλασική περίπτωση εδώ πέρα το του ότι δεν είχαμε εντοπίσει το εύθραυστο της κατάστασης και ακριβώς τονίζει το θέμα της αντοχής που πρέπει να υπάρχει. Αν υπήρχε ένα σύστημα στις χώρες αυτές υγείας, ίσως ε, να ήταν διαφορετική η κατάσταση σήμερα. Οπότε είναι ένα δίδαγμα στο οποίο πρέπει να επανέλθουμε και ε, θα γίνει. Δεύτερον, για την ε, πολιτική βούληση συμφωνώ με τον φίλο μας, τον Γκέρενς, πως χρειάζεται πραγματικά και προσπαθούμε να προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι. Ε, είχαμε πολύ σαφές ε, κατευθύνσεις από τους αρχηγούς ε, κρατών και κυβερνήσεων ακριβώς γιατί κάποιοι θεωρούσαμε πως δεν υπήρχε επαρκής πολιτική προσοχή. Και κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε η κυβέρνηση των ΙΠΑ. Ε, πόρους έχουν τα κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη προσπαθούν να δουν πώς θα τους αποστείλουν εκεί. Κάνουν τεράστια προσπάθεια, αλλά δεν έχουμε ακριβώς μία δομή... Ε, διοίκησης και ελέγχου. Προσπαθούμε ε, να ε, συντονίσουμε τον κόσμο, να πούμε αυτά είναι τα προβλήματα και κάντε το. Και αυτό το οποίο λάβαμε, η εντολή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν αυτή ακριβώς. Υπήρχε επιθυμία της ε, Κάθριν Μπέερ να δει το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. Αυτό ακριβώς ζητήσαμε. Δηλαδή, δώστε μας εντολή και το κάναμε 48 ώρες το σχέδιο. Το στείλαμε και βεβαίως ε, αφορά ατομικό εξοπλισμό προστασίας, ε, νοσοκομεία εκστρατείας, ε, αποκομιδή ασθενών, δυνατότητες μεταγωγικών κτλ. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά χρειάζεται και η στήριξή σας και το ψήφισμα βεβαίως του Στρασβούργου ήταν νομίζω πάρα πολύ καλή ε, όθηση και προς τα εκεί θα συνεχίσουμε. Προφανώς είμαστε σε επαφή με αυτούς οι οποίοι θα είναι στη συνάντηση στη Νέα Υόρκη. Τα είπε η κυρία Πρέσβη, στην Πέμπτη θα έχουμε τη συνάντηση και η Σαμάνθα επίσης θα πάει. Αλλά ε, προφανώς η Ευρώπη πρέπει να λάβει τις ευθύνες της. Για να είμαι ειλικρινής και εδώ πέρα μιλάω για την χρηματοδότηση, θεωρώ πως ε, είχαμε μείνει λίγο πίσω αλλά όχι τόσο πολύ. Κάποιος μίλησε για τον Μάρτιο, για τα πρώτα σημάδια. Η πρώτη εκταμείευση που κάναμε εμείς ήταν το Μάρτιο. 500.000, όχι πολλά. Αυτό βλέπαμε τότε. Και μετά τον Ιούνιο άλλα 2-3 εκατομμύρια. Μετά φτάσαμε στα 12. Μετά όταν είδαμε πώς είναι η κατάσταση, ο κύριος Πίμπαλξ ε, έδωσε 140 εκατομμύρια αμέσως χρησιμοποιώντας ε, το μέσο της κρίσης το λεγόμενο. Οπότε παρακολουθούμε την κατάσταση και τα νούμερα δεν είναι τόσο άσχημα. Τα κράτη-μέλη όλα κινητοποιούνται, είδα εγώ ένα έγγραφο πριν από δύο εβδομάδες, ε, που μιλούσε για 10 εκατομμύρια, σήμερα μιλάμε για 78 εκατομμύρια ήδη. Αυτή τη στιγμή συζητάω με τον DDA και τους υπόλοιπους φίλους ε, πώς μπορεί να δώσουμε άλλα 30 εκατομμύρια γιατί κάτι έχει γίνει. Αλλά κοιτάξτε, εγώ θέλω να κινούμαστε εμείς πιο γρήγορα γιατί η Ντεύκο κατά κανόνα ε, πηγαίνει, κινείται πιο μακροπρόθεσμα αλλά οπωσδήποτε θα βρεθούν και άλλα κονδύλια. Εάν πάμε τώρα στο αποθυματικό εκτάκτων αναγκών, μπορεί Ελπίζω να έχω τη στήριξή σας αν χρειαστεί κάτι τέτοιο. Ε, και οπωσδήποτε θα ξέρετε πού θα πάνε τα λεφτά. Για την κένωση προσωπικού και τα βαρέα μεταγωγικά. Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια να πείσουμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν. Χάρηκα που είδα το έγγραφο των Γάλλων συναδέλφων που έλεγε πως πρέπει να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση δεν είναι εύκολο γιατί σύμφωνα με τους κανόνες το κάθε κράτος μέλος έχει την ευθύνη για τους υπηκόους του και τους παίρνει τους εκενώνει κτλ. Το θέμα είναι πως έχουμε κράτη-μέλη που δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες, είναι μικρά. Έχουμε επίσης ε, στους γιατρούς χωρίς σύνορα προσωπικό από όλες τις χώρες ε, και πραγματικά δεν είναι δυνατόν να μισθώνουν αυτοί αμερικανικό αεροπλάνο για να κάνουν αεροδιακομιδές. Θα γράψω πάλι αύριο επιστολή στις αρχές ε, πολιτικής προστασίας ε, για να συνεννοηθούν στρατός και Υπουργεία Εξωτερικών για την οργάνωση των ε, αεροδιακομιδών. Θα είμαι στη Ρώμη τη Δευτέρα να τα κάνουμε όλα αυτά. Ευχαρίστω. Η πίεση από εσά καλοδεχούμενη γιατί δεν είναι εύκολο να συνεννοηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι αλλά νομίζω πως όλοι έχουν τις καλές προθέσεις. Μπορώ να σας δώσω για παραδείγματα πάνω σε, σε 130 διάφορες φούσκες κτλ. λοιπά, δεν χρειάζονται όλα αυτά. Όπως είπα λοιπόν πρέπει να υπάρξει με κάποια προσπάθεια εντός των θεσμικών οργάνων και βεβαίως να μην υπάρχει αλληλεπικάλυψη, να μην κάνουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Να βάρω, ο Ρίκ και όλοι οι υπόλοιποι που είναι εκεί επί τόπου πρέπει να έχουν τις δυνατότητες να δουλέψουν. Και εμείς να βοηθήσουμε αυτές τις δομές. Αυτό κάνουμε τώρα. Θα γίνει άλλο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα, υπό την Προεδρία της ε, Κρυσταλίνας ε, Γεωργίευα. Οπότε θα συνεργαστούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΚΟ, ο κύριος Βεύς. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να προσθέσω και εγώ δύο λόγια μετά από αυτά που είπε ο Διευθυντής της ΕΚΟ. Υπενθυμίζω ότι έχουμε να κάνουμε με την ανάπτυξη και θέλουμε η εκταμίευση να επιταχύνεται και ό,τι είχε προβλεφθεί να εκταμιευθεί, να εκταμιεύεται πράγματι θέλουμε έτσι και αλλιώς να γίνεται η εκταμίευση, ακόμα και αν δεν έχουν διασφαλιστεί κάποια προηγούμενα βήματα. Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε και το σεβασμό βέβαια των δημοσίων οικονομικών. Δεν γίνονται όλα αυτά σε βάρος του διαλόγου που έχουμε με τις χώρες μέλη για τη διαχείριση των πόρων. Και γιατί λέω ότι αυτά είναι σημαντικά, γιατί τα είπε πολύ σωστά ο πρέσβης προηγουμένως όλες οι χώρες στην περιοχή χάνουν 4% περίπου από την ανάπτυξή τους. Η Λιβερία ίσως και παραπάνω. Τα συζητάμε και με το συντονισμό του Διεθνούς Νομισματικού Τομείου, οπότε βρισκόμαστε στη λογική της διασφάλισης των εκταμιεύσεων, που θα χρησιμεύσουν σε τι θα χρησιμεύσουν να διασφαλίσουν τους μισθούς στον κοινωνικό τομέα, είτε πρόκειται για την υγεία, είτε πρόκειται για την εκπαίδευση όμως. Θα χρησιμεύσουν επίσης να πληρωθούν τομείς όπως η ασφάλεια. Έτσι κι αλλιώς ε, πολιτών, έτσι. Πρέπει οι δομές αυτές να εξακολουθούν να υπάρχουν. Με αυτή την οπτική λοιπόν δρούμε και εμείς και δίνουμε οικονομική στήριξη. Μια άλλη πτυχή σε αυτά που ανακοίνωσε ο Επίτροπος Πίβεταλτς είναι ότι θέλουμε από σήμερα να διασφαλίσουμε τη σύνδεση ανάμεσα στο ανθρωπιστικό και την ανάπτυξη. Πολλές φορές λείπει αυτός ο κρίκος. Έτσι λοιπόν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δρούν στον τομέα της υγείας, ανθρωπιστικής βοήθειας, ε, νερού κλπ θα στηριχθούν ακόμα και όταν η κρίση θα έχει περάσει σε ένα επόμενο στάδιο μείωσης ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί, αλλά θέλουμε να φροντίσουμε να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για να διασφαλιστεί αυτή η μετάβαση από την περίοδο κρίση την περίοδο μετά την κρίση. Και όπω ακούσαμε και από τι ΗΠΑ, ναι, υπάρχει συνεργασία με τι ΗΠΑ για το πρόγραμμα τη Αφρικανική Ένωση. Για να επανέλθω στι τρει χώρε, μιλήσαμε πολύ για τη Σιέρα Λεόνε και για την Λιβυρία. Στη Γουινέα η αλήθεια είναι ότι έχει σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι ο μεγαλύτερος δωρητής στον τομέα της υγείας. Με τα 11 εκατομμύρια λοιπόν εξακολουθούμε να δραστηριοποιούμε θα εκεί στον τομέα της υγείας και να διασφαλίζουμε ε, βασικές υπηρεσίες. Μακροπρόθεσμα, όπως ακούσαμε ήδη, πρέπει να συνεχίσουμε να ε, δουλεύουμε στη Δυτική Αφρική και να την κάνουμε πιο ανθεκτική όσον αφορά την υγεία. Για τις ερωτήσεις σας. Ναι, έχουμε ελαστικές διαδικασίες για τις τρεις αυτές χώρες. Ο δημοσιονομικός κανονισμός εφαρμόζεται με ελαστικότητα, τα έχουν πει αυτά οι αρμόδια από την Επιτροπή και ο Επίτροπος Σουμπίβελτς, και βέβαια το Αναπτυξιακό Ταμείο έχει μεγάλη σημασία. Όλες αυτές οι δράσεις γίνονται πραγματικότητα χάρη σε διατησίες. Όσο το ανδέκατο ΦΕΔ δεν έχει επικυρωθεί, εμεί δουλεύουμε με το Bridging Facility, την διάμεση διευκόλυνση δηλαδή. Οπότε τα χρήματα που εκταμιεύονται, πηγαίνουν καμιά φορά και στην ΕΚΟ, γίνονται βάσει διαιτησίας. Γιατί μερικές φορές έχουν προβληθεί χρήματα για άλλες χώρες, ακέ. Οπότε το Αναπτυξιακό Ταμείο αποτελεί προτεραιότητα αν θέλουμε το 2015 να μπορέσουμε να στηρίξουμε την αντιμετώπιση της κρίσης του ιού έμπολα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ο κύριος Στούπς από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Κυρίες και κύριοι του Κοινοβουλίου, έχω την τιμή να εκπροσωπώ σήμερα την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων και θα ήθελα από την αρχή να τονίσω τι είπε ο Κλάους προηγουμένως, ότι καθημερινά και κάθε ώρα σχεδόν είμαστε σε επαφή με τις υπηρεσίες και όσους ασχολούνται επιτόπου με την αντιμετώπιση της κρίσης. Δεν είναι όλοι εδώ βέβαια γιατί συνεργάζονται και με την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ και έχουν και δικές τους ευθύνες, ας πούμε, για να διασφαλιστεί ότι οι, αερογραμμές, οι δημόσιες αερογραμμές δεν θα ακυρώσουν τις πτήσεις τους από και προς τις χώρες της περιοχής. Καθώς λοιπόν κατανέμουμε την εργασία μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων και συντονιζόμαστε στενά, η δική μας υπηρεσία έχει ως προτεραιότητα το outreach καταρχήν προς την περιφέρεια, προς τις ε, πληττόμενες χώρες. Πολύ σύντομα οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών έλαβαν πολύ σκληρές αποφάσεις όπως κλείσιμο των συνόρων, ακυρώσεις πτήσεων. Εμείς όμως προσπαθήσαμε με όλα μας τα διπλωματικά μέσα να διευκολυνθεί να διευκολυνθούν αυτά τα άκαμπτα μέτρα και σήμερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί πολύ. Ας πούμε το αεροδρόμιο της Άκρα και του Ντακάρ έχει ανοίξει και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δύο αεροδρόμια για την εκένωση προσωπικού και για τη μεταφορά υλικού στις χώρες που πλήττονται από τον έμπολα. Αυτό λοιπόν άμεσα στις ενδιαφερόμενες χώρες που πρέπει να συνεχιστεί και στις γειτονικές. Δεύτερο μέτρο επιτόπιας, ε, επιτόπιου αποτελέσματος αφορά συγκεκριμένα τις χώρες της Ένωσης. Όπως είπε και ο Κλάους, τα όργανα της Ένωσης δεν έχουν πολλές δυνατότητες το πολύ που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποβάλουμε τα προβλήματα σε στρατιωτικούς και πολιτικούς εκπροσώπους επιτόπου. Τι Ίσως να θεωρήσετε τολμηρό ότι μέχρι τώρα πρέπει να πω είδαμε κάποιους δισταγμούς από τα κράτη-μέλη. Δεν ανέλαβαν καθαρά την ευθύνη της μεταφοράς ιατρικού υλικού και προσωπικού. Γνωρίζουμε ότι είναι κατεπήγον το θέμα και ποιες είναι οι ανάγκες. Όπως μας είπε και ο Διευθυντής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και πολλές φορές το θέμα, το πρόβλημα έγκυται στους πολιτικούς ηγέτες. Και δύο τελευταία. Το προσωπικό. Όσοι δολοφονήθηκαν στη Γουινέα Μπισάου. Ήταν κάτι που το ανέλαβε συνολικά η Ένωση και είναι σημαντικό νομίζω το outreach που σας έλεγα, το outreach. Για να φανεί και στις ενδιαφερόμενες χώρες ότι υπάρχει πολιτική θέληση. Thank you. I just have um, two colleagues want to make quick Δύο συνάδελφοι θέλουν κάτι να πούνε και μετά επισκέπτες μας αν θέλουν να αντιδράσουν σε αυτά που άκουσαν είτε από τους ευρωβουλευτές είτε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ο κύριος Δεμέρα. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Οι γιατροί χωρίς σύνορα λένε ότι η επιδημία έχει ξεφύγει. Λένε ξεκάθαρα ότι αυξάνονται τα θύματα κάθε εβδομάδα. Μας λέει επίσης ότι δεν υπάρχει προηγούμενο όντως. Άρα βρισκόμαστε μπρος σε μια έκτακτη κατάσταση επίγουσας ανάγκης. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει απομόνωση, θεραπεία και εκένωση. Αυτά τα τρία. Και χρειάζεται κάποιος ο οποίος θα συντονίζει, θα ελέγχει. Έχω πολλά σχόλια, αλλά προσπαθώ να σας τα πω σύντομα, μια που μου είπατε να βιαστώ. Η πρόταση του Ενρίκε Γκερέρο πιστεύω ότι είναι καλή και ενδιαφέρουσα. Στην Ισπανία έχουμε τρεις διορθών, όχι δύο περιπτώσεις, τρεις θύματα. Ο πρέσβης τώρα από τις χώρες ΑΚΕ. Είναι ενδιαφέρουσα η πρότασή του, αλλά θέλω να σας πω ότι πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η Προεδρία τελειώνει τον Δεκέμβριο και ίσως να μπορούμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια να αποφασίσουμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στο έμπολα. Σύντομα κύριε Γκόρενς. Ναι, ναι κύριε Πρόεδρε. Αυτά που είπε ο κύριος Σάρενσεν και εκπρόσωπος της ΕΑΣ με ταρακούνησαν κάπως. Όντως τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους το Συμβούλιο πρέπει να το καλούμε σε κάθε συνεδρίασή μας και να έρχεται και να λογοδοτεί για το τι κάνουν οι χώρες μέλη για αυτή την τόσο λεπτή και σοβαρή περίπτωση. Σιωπά κατά τη διάρκεια όλης της θητείας αυτής. Εγώ θέλω να έρθει το Συμβούλιο και να μας πει πώς θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ευχαριστούμε. Ναι, θα στείλουμε μια επιστολή πιστεύω στον πρόεδρο του Συμβουλίου και για το συντονισμό και γι' αυτό. Ωραία. Οι προσκεκλημένοι μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο βέβαια. Έχετε κάτι να απαντήσετε. Δύο λεπτά. Ο κύριος Πρέσβης μήπως. Για το θέμα της ε, τριμερούς απομόνωσης, βοηθάει στο να συνειδητοποιήσει ο κόσμος περί ως πρόκειται. Τώρα το έχουν όλοι συνειδητοποιήσει. Όταν ε, άρχισε ο ιός έμπολα να μεταδίδεται, ο κόσμος τον αρνιόταν. Αρνιόταν να πάρει θεραπεία. Αυτό έχει αλλάξει. Το δεύτερο όφελος από το τρίμερο αυτό απομόνωσης ήταν ότι δείξαμε την αποφασιστικότητά μας προς τον ε, υπόλοιπο κόσμο. Ότι δηλαδή παίρνουμε πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και τρίτον, η τρίτη επίπτωση είναι ότι ο κόσμος είναι ενημερωμένος και για τα θέματα δημόσιας υγείας, δηλαδή ότι πρέπει να καθαρίζει, πώς πρέπει να καθαρίζει, ότι συνειδητοποιημένα πρέπει να προσέχει τι τρώει, πώς το τρώει, για να είναι ασφαλές το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Ήταν η εποχή που είχαμε και την ε, ελονοσία και την ε, χολέρα την ίδια εποχή με την ε, έκρηξη αυτή του ιού έμπολα. Οπότε το θέμα της συνδυτοποίησης πέρασε στην πρώτη γραμμή. Τώρα κατά πόσο η επιδημία αυτή επηρεάζει τους αναπτυξιακούς στόχους, ναι, όπως είπε και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ναι, πλήττεται έτσι και η δικιά μας αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε με τους αναπτυξιακούς στόχους. Παραμένουμε στα ίδια επίπεδα. Δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα ή απειρολάχιστη. Η πίεση είναι μεγάλη για το υγειονομικό προσωπικό που πρέπει να πηγαίνει να βοηθήσει στις χώρες που πλήττονται. Γιατί βλέπετε οι άλλες χώρες κλείνουν τα λιμάνια τους στα σκάφη που έρχονται από τις χώρες που έχουν πληγεί. Άρα δυσκολεύεται αυτή η επαφή, αυτό το εμπόριο πρέπει και αυτές οι χώρες να πιστούν και να καταλάβουν ότι όταν έρχονται εμπορεύματα ή πλοία από τις χώρες που έχουν τον ιό έβολο δεν σημαίνει ότι αυτόματα μολύνονται κιόλα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε άλλος. Κανείς, ε, γιατροί χωρίς σύνορα. Σύντομα, τι μήνυμα έχετε να μας μεταφέρετε. Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε Τώρα είναι για το κατεπήγον, έτσι, για την έκτακτη κατάσταση. Δεν ναι, θέλω απλώ να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Όντω έχουμε έναν υγειονομικό υπάλληλο μέλο που έχουμε που έχει μολυνθεί. Βλέπετε και με τον προσωπικό, το, ε, την προστασία την προσωπική ε, υπάρχει κίνδυνος παρόλο που φροντίζουμε και να χρησιμοποιούμε χλωρίνη και ο ένας να ελέγχει τον εξοπλισμό του άλλου ώστε να μην παραβλέψει κανείς τίποτα στον ε, εξοπλισμό του προστασίας. Πάντως δεν υπάρχει θεραπεία ακόμα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φροντίσουμε για την απομόνωση, ενυδάτωση και λύση άλλων υγειονομικών προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν. Έχουμε 40 με 50 μονάδες κλινών. Στη Μονραβία έχουμε 200, ενώ θα θέλαμε 400. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την ανάληψη κινδύνου από πλευράς του υγειονομικού προσωπικού. Ποτέ δεν είχαμε πάντως τέτοια μονάδα απομόνωσης. Γιατί κινδυνεύει το προσωπικό, γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση να δέχεται όλο και περισσότερα, γιατί δεν υπάρχουν αρκετές μονάδες ολόκληρη τη χώρα, οπότε ταξιδεύει ο κόσμος από την Μονοραβία για να πάει σε αυτές τις δυο τρει μονάδες που είναι ανοιχτέ ακόμα. Ένα από τα μαθήματα πάντως που παίρνουμε από την παρέμβαση την τωρινή αλλά και τι παλιότερε είναι το θέμα της αξιωτικής παρέμβασης. Όχι, εμείς ζητάμε προστασία των πολιτών ε, από Υπουργεία Υγείας. Λέμε ότι η προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική και να είναι σαφές το ποιος δίνει τις εντολές. Οπότε γι' αυτό το θέμα μερικές φορές η στρατιωτική είναι μια καλή λύση γιατί έχουν τη συνήθεια να δίνουν εντολές. Γιατί ακόμα και στα κοινοτικά θεραπευτικά κέντρα και εκεί χρειάζονται αυστηρές προδιαγραφές. Αλλιώς μπορεί να μπερδέψεις τους ασθενούντες από ελονοσία με εκείνους που έχουν έμπολα. Πρέπει να γίνεται διαχωρισμός αυστηρός και η οργάνωση να είναι πάρα πολύ καλή. Και στα κέντρα λοιπόν αυτά για τον έμπολα χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Όλα αυτά βέβαια υπογραμμίζουν και πάλι το θέμα της ταχύτητας. Η ταχύτητα είναι ένα θέμα, για τόσο πιο πολύ περιμένουμε, τόσο περισσότερο ο ιός κινδυνεύει να μεταδοθεί και να πάει στις γειτονικές χώρες. Από τις τρεις που πλήττονται ήδη. Και τόσο πιο δύσκολο θα είναι να διαχειριστούμε αυτά τα μεγάλα θεραπευτικά κέντρα τα οποία θα πιέζονται συνεχώς να δεχτούν όλο και περισσότερους ασθενείς. Συνεπώς η ταχύτητα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για να τελειώσω εγώ γρήγορα όπως μου είπατε αλλά και για να αντιμετωπίσουμε τον ιό. Ωραία. Πέντε λεφτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας. Κάτι επίγον πρέπει να ακούσουμε από τους άλλους μας προσκεκλημένους. Όχι. Α, ναι, παρακαλώ. Πολύ σύντομα για το θέμα του... της ταχύτητας. 44 μονάδες έχουν σχεδιαστεί στις τρεις ή μάλλον πιο στα στις πέντε χώρες. 20 είναι έτοιμες. Αυτό τι σημαίνει. Μετά το κυκλώνα στις Φιλιππίνες είχαμε 150 μονάδες που πήγαν. Άρα προφανώς και είμαστε πολύ πίσω. Προστασία του πολίτη, οργανώσεις δηλαδή που ασχολούνται με αυτό το θέμα ή εθνικές στρατιωτικές αρχές επίσης πρέπει να συμμετέχουν. Αν δείτε τα διάφορα γραφήματα που λένε κάνουν την πρόβλεψη φαίνεται ότι θα έχουμε χιλιάδες περιπτώσεις κάθε εβδομάδα. Έχουμε δύο κυβερνήσεις που περιμένουν να έρθουν ομάδες, που ελπίζουν να έρθουν ομάδες. Πρέπει να είναι συλλογική προσπάθεια. Και να απαντήσω και σε μια ερώτηση. Αν έχουν ανοσία οι ασθενείς που έχουν ήδη μάλλον ασθενείς και έχουν θεραπευτεί, έχουν μεγάλη ανοσία και χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν με διάφορους τρόπους να ανθαρρύνουν τον κόσμο, να ζητήσει βοήθεια κλπ. κλπ. Πρόεδρος, το θέμα της εκένωσης είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί που πηγαίνουν εκεί πρέπει να νιώθουν ότι με ασφάλεια θα επιστρέψουν στις χώρες τους αν νοσήσουν. Και υπόθηκαν αυτά και σε άλλες συναντήσεις που έγιναν. Άκουσα την πρόταση του κύριου Γκερέρο. Πού τη στήριξαν. Τη στηρίζουν νομίζω όλοι οι συνάδελφοι. Οπότε λέω να ετοιμάσουμε μια επιστολή και να τη στείλουμε στην Προεδρία του Συμβουλίου αμέσως και στην είπα το εκπρόσωπο. Ίσως με αντίγραφο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της εκένωσης. Θα το συζητήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δούμε τελικά ποιος θα πάρει την απόφαση. Αλλά σίγουρα πρέπει να τη στείλουμε αυτή την επιστολή. Και έχουμε βέβαια και την έκθεσή μας, η οποία θα αντιμετωπίσει και το θέμα το μακροπρόθεσμο. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συνάντηση. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος. Ακυρώνεται η συνεδρίαση της Επιτροπής μας για την επόμενη εβδομάδα λόγω των ακροασών. Θα τα μάθετε από τους συντονιστές σας. Δευτέρα και Τρίτη βράδυ έχουμε δύο επιτρόπους. Θα τα ακούσετε από τους συντονιστές σας. Και πάλι ευχαριστώ. Έλειξε η συνεδρίαση. I should have said we have this afternoon, of course, at 3 o'clock the meeting. We resume at 3 o'clock with climate change and votes and then Sakharov Prize. Απόγευμα τα ξαναλέμε, κλιματική αλλαγή, Ζαχάροφ, ψηφοφορίες κτλ.